Okay, let us begin by... Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρώτο σημείο. Έγκριση της ημερήσια διάταξης. Να σας ενημερώσω για την εξής αλλαγή που έγινε στο σχέδιο ημερήσια διάταξης. Το σημείο 14 αναβάλλεται και το σημείο 4 θα το συζητήσουμε μετά το σημείο 12. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θεωρώ ότι η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί όπως τροποποιήθηκε. Να σας ενημερώσω επίσης ότι η συνεδρίασή μας είναι δημόσια, μεταδίδεται στο διαδίκτυο, εκτός από τα σημεία που θα συζητηθούν και κλεισμένων των θυρών. Και να σας ενημερώσω ότι όλες οι χρονοθυρίδες είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να αλλάξουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας. Σημείο 2. Δεν έχω ανακοινώσει. Οπότε μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 3. Άρθρο 42, επικουρικότητα. Σημειώστε παρακαλώ. το σημείο αυτό και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 5. Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Ο λόγος στον εισηγητή μας, τον κύριο Μαστάλκα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Λίγα λόγια να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο καρκίνος είναι ο σημαντικότερος και συχνότερος λόγος θανάτου, ιδίως όσον αφορά τις ασθένειες που προέρχονται από το χώρο εργασίας. Και ως εισηγητής για την οδηγία αυτή με την οποία ε, τροποποιείται η οδηγία 37 του 2004 σε σχέση με την προστασία των εργαζομένων από τους μεταλλοξεργάνους και καταρκυνογόνους ε, παράγοντες. Εγώ θέλω να δηλώσω την πλήρη υποστήριξή μου προς τις προθέσεις της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ορίζονται λοιπόν οριακές τιμές για το κάδμιο, τις ανόργανες ενώσεις του, το αυρίλιο, τις ε, ε ενώσεις του, το αρσενικό, τη φορμαλδεΐδη και την 4-4 μεθυλοαναλίνη. Στην πρόταση οδηγίας αναφέρεται ότι η καλύτερη προστασία από τους κατοικογόνους και μεταξυβελογόνους παράγοντες ε, θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της κατάστασης, θα προστατευτούν πάνω από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι και θα ε, μειωθούν 20, κατά 22.000 οι περιπτώσεις ε, καρκίνου που σχετίζονται με την εργασία. Έχω κάνει κάποιες τροπολογίες σε σχέση με την καλύτερη προστασία, κάποιες προσθήκες ουσιών στον κατάλογο βάσει των επιστημονικών στοιχείων που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας. Επίσης, προτείνω τη μείωση της μεταβατικής περίοδου εφαρμογής των ε, οριακών τιμών για τις ουσίες αυτές. Ελπίζω να τύχει η πρότασή μου αυτή της υποστήριξής σας. Τροπολογίες μπορείτε να υποβάλλετε έως τις 7 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ και προσβλέπω στη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Κύριε Ζώμητη έχει το λόγο. Well, I believe that one needs Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα τον εισηγητή για τη δουλειά του. Συμφωνούμε σίγουρα ότι το να διασφαλίζουμε πω οι εργαζόμενοι δεν θα <clears throat> εκτίθενται σε τέτοιου είδου παράγοντες είναι απόλυτος απαραίτητο. Μειώσαμε καταρχήν τις ουσίες σε 21 και τώρα ε, συζητάμε τα όρια για περισσότερες ουσίες. Τα χημικές ουσίες για τις οποίες γίνεται λόγος δεν προκαλούν απλώς καρκίνο, που είναι ήδη πολύ σοβαρό, αλλά δημιουργούν και άλλου τύπου προβλήματα όπως ε, στο αναπνευστικό σύστημα και στο νευρικό σύστημα. Πρόκειται για χημική, χημικούς παράγοντες που είναι παρόντες ε, στα εργαστήρια, στον τομέα των ηλεκτρονικών, στην οικοδομή, ε, στον τομέα της υγείας, στα πλαστικά, στην επεξεργασία αποβλήτων και αλλού. Χρειάζεται λοιπόν να προλάβουμε τους κινδύνους. Σε ό,τι αφορά τη Μάλτα, μικρή χώρα, αλλά παρόλα αυτά έχουμε 2.000 νέες περιπτώσεις καρκίνου το χρόνο και περίπου 1.000 θανάτους ετησίως από καρκίνο. Πρέπει να καταπολεμούμε τον καρκίνο συνεχώς μέσω της έρευνας, αλλά και στον τόπο εργασίας διότι οι εργαζόμενοι παίρνουν πολλές ώρες από τη ζωή τους εκεί και ο καρκίνη εξαιτία παραγόντων στο περιβάλλον εργασία είναι πολύ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 22.000 συνολικά ετησίως κατέτος. Θα βελτιώσουμε έτσι τη ζωή ενό εκατομμυρίου, ε, εργαζομένων. Ε, συμφωνώ με τον εισηγητή σε ένα μόνο σημείο όμως θα πρέπει να παραμείνουμε στην πρόταση τη Κομισιόν και να μην την τροποποιήσουμε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο και την εισαγωγή νέων ορίων. Το λέω διότι η πρόταση της Κομισιόν βασίζεται ήδη σε διαβούλευση με τους επιστημονικούς φορείς, τους εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργοδοτών κλπ. Είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα, οπότε θα πρέπει να το χειριστούμε με τον ορθότερο δυνατό ε, τεχνικό και επιστημονικό τρόπο. Η Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην, ε, στο χώρο εργασία βρίσκεται σε διαβούλευση μαζί μα και με την Κομισιόν και το ίδιο και η κοινωνική εταίρη. Ε, μία πρόταση του εισηγητή, δηλαδή να εξετάσουμε περισσότερο το θέμα του ποια είναι τα πιο κατάλληλα όρια έκθεσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά και θα δεχτώ την τροπολογία, αλλά θα προσθέσω πως πρέπει να γίνει περισσότερο ερευνητικό έργο ε, με όλους τους αρμόδιους φορείς. Όλα αυτά όμως δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε πρόσθετα διοικητικά βάρη. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, would the Commission wish to take the floor? Commission? Doesn't seem to be the... Όχι, δεν φαίνεται να θέλει το λόγο. Προθεσμία για τις τροπολογίες 7 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Κλείνουμε αυτό το θέμα. Και περνάμε στο σημείο 6. Ε, διαφάνεια και βιωσιμότητα του συστήματος εκτίμησης κινδύνου στην τροφιμική, αλυσίδα. Και πάρει ο κ. Μαστάλκα. Ευχαριστώ, συναδελφοί, για τη συζήτηση στο προηγούμενο θέμα. Αυτή η πρόταση δεν θα είναι τόσο απλή όμως. Είναι πιο επίμαχη. Η πρόταση της Κομισιόν ήδη ήταν επίμαχη. Η υπόθεση της γλυφοσάτης δημιούργησε πολλές αντιδράσεις και αιτήματα πλευράς των πολιτών υποπίεση κινδύνου βέβαια, το γνωρίζουμε αυτό. Παρ' όλα αυτά, η πρόταση αυτή πιστεύω πως δεν είναι πλήρης. Ε, δεν έγινε αξιολόγηση επιπτώσεων και το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιεστικό. Δεν νομίζω θα καταφέρουμε να τελειώσουμε κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μας. Και αν το κάνουμε, η ποιότητα του νομοθετικού κειμένου δεν θα είναι η κατάλληλη. Η πρόταση κομισιών είναι το πρώτο σωστό βήμα. Για παράδειγμα, αυτόματη αποκάλυψη δεδομένων σε μορφή που μπορεί να αναγνωστεί από μηχανές, ενημέρωση <clears throat> των ε, μερών και η ανανέωση της σύνθεσης της Εύσα Όμως, η Κομισιόν δεν εξασφαλίζει με αυτή την πρόταση τον μέγιστο βαθμό διαφάνεια. Για παράδειγμα, υπάρχει μια πρόταση σύμφωνα με την οποία τα επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικέ μελέτε δημοσιοποιούνται όταν ε, ε, κατατίθενται αιτήματα για μη γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν προστατεύεται η πνευματική του ιδιοκτησία ενώ των μελετών και των δεδομένων. Όμως υπάρχουν τόσο πολλές εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα που τελικά πλήττεται η διαφάνεια. Δεν θα πρέπει Επίση να λαμβάνει υπόψη όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από την σύμβαση του άρχου. όπως λέει η Κομισιόν. Ποιο επίση θα χρηματοδοτήσει την επιβεβαίωση την, αυτών των μελετών. Η Κομισιόν λέει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να γίνει με κρατικά κονδύλια. Αυτό σημαίνει τελικά όπω το καταλαβαίνω εγώ, ότι οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν τι εταιρείε. Έχω 78 τροπολογίες στις προτάσεις Κομισιόν. Η διαφάνεια είναι σημείο κλειδί. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να είναι δυνατόν να αποφεύγεται η δημοσίευση, η δημοσιοποίηση των πληροφοριών όταν κινδυνεύει το περιβάλλον ή η δημόσια υγεία. Μόνο έτσι μπορούμε να τηρήσουμε την αρχή της προφύλαξης. Το... Η νομική, η ασφάλεια δικαίου θα πρέπει να εξασφαλιστεί. Το απόρριτο και η εμπιστευτικότητα θα πρέπει να οριστούν όσο πιο στενά γίνεται. Η έγκαιρη δημοσιοποίηση πληροφοριών και μελετών είναι σημείο κλειδί. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα στη συζήτηση αυτή τη νομοδοτηση. Θα δυσκολευτούμε να βρούμε ισορροπημένε λύσεις. Περιμένω όμω τις νόμες, τη γνώμη σα και τις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε κυρία Ντελβό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κύριος Γκάσπαρα είναι σκιώδη, ζητεί συγγνώμη που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Θα διαβάσω τη δήλωση του. Η πρόταση της Επιτροπής για τη διαφάνεια και την βιωσιμότητα της μελέτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την διατροφική αλυσίδα αποτελεί ένα ζήτημα ύψης της σημασίας που αφορά την υγεία καθώς και την ευημερία των πολιτών και την προστασία των καταναλωτών, των ζώων και του περιβάλλοντος. Η πρόταση μας δίνει τη δυνατότητα να αναθεωρήσουμε τη λειτουργία της ΕΦΣΑ, βελτιστοποιώντας την διάφρωση της και χρειαζόμαστε φυσικά και ανθρώπινους πόρους, έτσι ώστε ο οργανισμός να είναι πιο αποδοτικός ως προς τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί και να είναι και πιο διαφων... διαφανής. Πρόκειται για θέματα ύψης της σημασίας, γι' αυτό θα πρέπει να εγγυηθούμε ώστε τα κατάλληλα και επαρκή μέσα διατίθενται στην ΕΦΣΑ έτσι ώστε να μπορεί να προβεί σε ελέγχους, σε ελέγχους υψηλής ε, ποιότητας σε σχέση με τους ενδεχόμενους κινδύνους στη διατροφική αλυσίδα. Δυστυχώς, τώρα τελευταία, δεχτήκαμε, μάλλον επισκεφθήκαμε την ΕΦΣΑ στην Πάρμα, μία αντιπροσωπεία την επισκέφθηκε. Υπάρχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες και περιορισμένο προσωπικό, κάτι το οποίο φύγει την ε, αυτονομία της όσον αφορά την, ε, τις διάφορες έρευνες για τοξικές ουσίες στη διατροφική αλυσίδα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό 178 κάθετος 2002 έτσι ώστε να ενισχύσουμε το σύστημα πιστοποίησης και αδειοδότησης της ΕΦΣΑ. Επίσης θα πρέπει να είναι βασικό μας μέλημα η ασφάλεια τροφίμων και να υπάρχουν και οι συναφείς εγγύσεις. Μόνο κατά αυτό τον τρόπο η βιομηχανία τροφίμων της Ευρώπης θα θεωρηθεί ορόσημο για καλή ποιότητα και ασφάλεια. Ζητούμε περισσότερες επενδύσεις στην ΕΦΣΑ, επενδύσεις ώστε να έχουμε τις υψηλότερες προδιαγραφές για την ασφάλεια τροφίμων και επίσης να μην επηρεάσει το οργανισμός από τους ιδιωτικούς ε, φορείς και μεγάλους οργανισμούς. Εδώ γίνεται μία αναφορά στα έγγραφα της Μονσάντο. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια για τους πολίτες και καλή διαχείριση διανομής δεδομένων, έτσι ώστε να υπάρχει σωστή ανταγωνιστικότητα στην αγορά, προωθώντας την καινοτομία και προωθώντας επίσης και την πνευματική ιδιοκτησία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα νομικά μέτρα έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η υγεία και η ευημερία των πολιτών. Όταν μιλάμε για την ε, υγεία των πολιτών ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πρωταρχικό μας μέλημα σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δρούν σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει λοιπόν η ΕΦΣΑ να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και της διαχείρισης κινδύνου. Και αυτό μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής ε, της ΕΦΣΑ. Ο κύριος ε, Ράτζεφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, βασικό μας μέλημα σε σχέση με τον κανονισμό για την ε, διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων αφορά την διασφάλιση μεγαλύτερης ε, διαφάνειας καλύτερης ε, και καλύτερης διαφάνειας ως προς τις επιστημονικές μελέτες, έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητες αυτές οι μελέτες και να προωθήσουν την επιστημονική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και να υπάρχει και καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σε σχέση με την αποτίμηση κινδύνου. Ένα από τα βασικά προβλήματα των πολιτών είναι ότι η αξιολόγηση κινδύνου στη διατροφική αλυσίδα, οι αξιολογήσεις αυτές ε, δεν είναι αξιόπιστες και ασφαλείς. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόβλημα της γλυφοσάτης. Εδώ και μήνες για πολλούς μήνες δεν γνωρίζαμε κατά πόσο η αδειοδότηση θα παραταθεί για ποια χρονική περίοδο και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση καθώς και σε αρκετές άλλες υπάρχει έλλειψη επαρκών και αξιόπιστων πληροφοριών σε σχέση με τους κινδύνους που απορρέουν από ορισμένες ουσίες ή προϊόντα. Όταν λοιπόν αυτές οι ουσίες έρχονται σε άμεση επαφή με την αλυσίδα τροφίμων, θα πρέπει να αποτιμήσουμε αυτούς τους κινδύνους επαρκώς, γιατί πλήττουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, τη σταθερότητα της αγοράς, της επενδύσεις και ούτω καθεξής. Το ρυθμιστικό λοιπόν πλαίσιο για την ασφάλεια τροφίμων θα πρέπει να ε, εγγυάται την σωστή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων σε σχέση με την αποτίμηση κινδύνων. Η πρόταση της Επιτροπής είναι απόλυτα απαραίτητη και ελπίζω οι πολίτες και οι καταναλωτές να ξέρουν ότι βασίζονται σε σωστές μελέτες σε σχέση με την ύπαρξη κινδύνων στην αλυσίδα τροφίμων. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τα μέτρα που θα προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα χωρίς όμως να γίνουν ε, ιδιαίτερα επιβαρυντικές αυτές οι διαδικασίες στον τομέα των ε, εμπειρογνωμόνων αλλά και των επιχειρήσεων. Ευχαριστούμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της DG τον κύριο Σκάνερ. Θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο εν γέννη για το πολύ επικοδομητικό του έργο σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν. Χρήσιμο είναι να σας θυμίσω το υπόβαθρο. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την απαγόρευση της γλυφωσάτης, όπου η Κομισιόν απάντησε ότι κατανοεί τις ανισοχίες των πολιτών για το γεγονός ότι το ενωσιακό πλαίσιο θα πρέπει να ενισχυθεί και ότι, ότι υπάρχει μια θεμελιώδης ανάγκη να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα ε, αξιολόγησης κινδύνου. Ταυτόχρονα, μέσω της, ε, του ελέγχου καταλληλότητας που έγινε για, το γενικό, για την Γενική Νομοθεσία για τα Τρόφιμα, η Κομισιόν αναγνώρισε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι στην Ευρώπη έχουμε τα πλέον ασφαλή τρόφιμα στον κόσμο. Χρειάζεται πολλή δουλειά βεβαίω. Και ε, η δουλειά μας έχει στεφθεί με επιτυχία, αλλά για να διατηρηθεί αυτή η επιτυχία πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν υποβάλαμε τη σχετική πρόταση. Κατανοώ λοιπόν ότι υπάρχουν πολλοί ευρωβουλευτές που ανησυχούν για το γεγονός ότι δεν υπήρξε μελέτη αντικτύπου, και εκφράστηκαν τέτοιε απόψει και εδώ, στην Επιτροπή σας. Η Κομισιόν όμως θέλει να τονίσει ότι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα συγκεκριμένο τμήμα του συστήματος τροφίμων. Το, το σύστημα που, που σχετίζεται με την αξιολόγηση κινδύνου και την διάσταση συγκεκριμένα της διαφάνειας αυτής της διαδικασίας. Και σε αυτό το πλαίσιο η πρότασή μας αποσκοπεί στο να εξασφαλιστεί ότι η ΕΦΣΑ θα έχει περισσότερα μέσα και νομιμοποίηση στην ε, εκτέλεση των καθηκόντων της. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ΕΦΣΑ θα λογοδοτεί στους Ευρωπαίους πολίτες με δημοκρατικό τρόπο. Και αυτό βεβαίως περιλαμβάνει και το θεμελιώδη ρόλο του Κοινοβουλίου. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε τις διατήξεις τις διατάξεις για τη δημοσιοποίηση όλων των μελετών και των δεδομένων που υποστηρίζουν αιτήσει εταιρεών ε, σχετικά με την έγκριση συγκεκριμένων ουσιών και πολύ συγκεκριμένα ακόμη περισσότερο στα φυτοφάρμακα και τα ζυζανιοκτώνα. Και βασικό στοιχείο της πρότασης της Κομισιόν είναι ότι πλέον απαιτείται η έγκαιρη αποκάλυψη, δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών για να εξασφαλιστεί η μέγιστη διαφάνεια. Και σκοπό μα είναι οι ετούντε όταν υποβάλλουν τι αιτήσει του, αιτήσει έγκριση συγκεκριμένων ουσιών, να υποβάλλουν και συνοδευτικέ μελέτε υποστηρικτικές οι οποίε θα δημοσιοποιούνται σε όλου του εμπλεκόμενου και ενδιαφερόμενου φορεί συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ε, προστασία και των θεμητών συμφερόντων των ε, κλάδων της οικονομίας μας και της καινοτομίας εν γέννη στην Ευρώπη. Ο κόσμος είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικός ε, και ο κλάδος των τροφίμων είναι πολύ ανταγωνιστικός και ε, βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας είναι η καινοτομία του, του κλάδου της οικονομίας αυτής. Επενδύονται τεράστια ποσά προκειμένου να εξασφαλίζεται η παραγωγή αλλά και η διάθεση στην αγορά καινοτόμων και ασφαλών προϊόντων στον κόσμο. Αυτό βεβαίω έχει πάρα πολλά ωφέλη στην Ευρώπη, ε, και τη απασχόληση. Άρα, παράλληλα με την έγκαιρη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, κάνουμε κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστούν τα θεμητά, τονίζω το θεμητά, συμφέροντα των εταιριών μας, των επιχειρήσεών μας όσον αφορά το απόρριτο, το επιχειρηματικό, τα εμπορικά μυστικά κτλ. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν ε, καταρτήσαμε έναν εξαντλητικό θετικό κατάλογο πληροφοριών ε, που πρέπει να δημοσιοποιούνται και έναν κατάλογο πληροφοριών που ε, παραμένουν εμπιστευτικές. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, εσείς προτείνατε να δημιουργηθεί ένας θετικός και ένας αρνητικός κατάλογος. Εμείς όμως έχουμε πολύ μεγάλο, μεγάλη εμπειρία στην DG Sante για όλα τα είδη προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, φάρμακα, τρόφιμα και πρέπει να σας πω ότι θετικοί κατάλογοι δεν συνεπάρχουν συνήθως με αρνητικούς καταλόγους. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν επιλέξαμε να καταρτήσουμε έναν θετικό κατάλογο ε, ουσιών. Εξασφαλίζουμε λοιπόν ότι τα ε, δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας και αποκλειστικότητας δεδομένων θα προστατεύονται υπέρ των πολιτών μας, της απασχόλησης Τη ε, καινοτομία και του καινοτόμου χαρακτήρα του κλάδου των τροφίμων. Επίση, προβλέπουμε, και αυτό είναι πολύ σημαντική διάσταση για του πολίτε, ότι θα υπάρχει δημόσια διαβούλευση έπειτα, ε, όσον αφορά τι ε, ε, μελέτες, ώστε η ΕΦΣΑ να έχει στη διάθεσή τη όλε τι απαραίτητε πληροφορίε για τι αξιολογήσει κινδύνου που θα διεξάγει. Και προκειμένου να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία, έχουμε προτείνει και ένα σύστημα κοινοποίηση των μελετών της Κομισιόν, ώστε όλοι να γνωρίζουν τα δεδομένα επί των οποίων θα εργάζεται η ΕΦΣΑ. Και ξαναλέω, αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη διάσταση της διαφάνειας. Άλλη πρόταση που επίσης είναι σημαντική στο πλαίσιο της καινοτομία και ιδίω όσον αφορά τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το εξή. Προβλέπεται η δυνατότητα εμ, συνάντηση πριν από την υποβολή μιας αίτηση, ώστε η ΕΦΣΑ να δίνει συμβουλές στους ετούντε για το πώς μπορούν να ε, εκπληρώσουν τις ε, απαιτήσεις, τις υποχρεώσει τους. Γνωρίζουμε ότι εκεί κάποιοι ε, φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των ετούντων και της ασφάλειας των τροφίμων. Από την άποψη δηλαδή ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια μεροληψία υπέρ του ετούντα. Εμείς όμως θεωρούμε ότι ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται και μετριάζεται. Και αυτό μέσω της ε, ιδιαίτερης ε, προσοχής που δίνουμε στη διαφάνεια και όσον αφορά αυτές τις συναντήσεις πριν από την υποβολή αίτησης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις μικρόμεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το ρυθμιστικό μας πλαίσιο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει στον τομέα τη ασφάλεια τροφίμων. Αναγνωρίζουμε ότι προφανώ είναι πολύ επιβαρυντικές ε, αυτέ οι διαδικασίε για μικρομεσαίες επιχειρήσει. Δεν είναι, δεν είναι συχνά πρόβλημα για τι μεγάλε εταιρείε τροφίμων, αλλά είναι πρόβλημα για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει και αυτέ θέλουμε να διευκολύνουμε. Χωρί βεβαίω να θέτουμε σε κίνδυνο καθόλου την ασφάλεια των τροφίμων. Μια άλλη διάσταση που σχετίζεται με το έργο και τη διακυβέρνηση του έργου αυτού είναι το εξή. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι ο ΕΦΣΑ θα έχει στη διάθεσή του ε, την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη. Το εύρος των εργασιών που καλύπτει ο ΕΦΣΑ είναι τεράστιο. Ε, αφορά ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχει ο ΕΦΣΑ στη διάθεσή του την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη, την καλύτερη δυνατή επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη ε, στην Ευρώπη. Αυτό βεβαίως πάντοτε με ανεξαρτησία, αμεροληψία κτλ. κτλ χωρίς να υπάρχουν σύγκρουση συμφερόντων. Και εδώ δηλαδή ανταποκρινόμαστε στο αίτημα για υψηλότερη διαφάνεια, ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία και μη σα πω να βελτιωθεί κιόλα. Και στο πλαίσιο λοιπόν τη διακυβέρνηση προτείνουμε τα κράτη-μέλη να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή και εμπλοκή στην διασπορά των ε, πληροφοριών ε, σε σχέση με την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη ε, και με την πρόταση συγκεκριμένων επιστημόνων. Και εδώ προσπαθήσαμε πάλι να εξισορροπήσουμε την επιστημονική επάρκεια και τη διαθεσιμότητα των επιστημονικών ε, πληροφοριών χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει καμία σκιά, χωρίς να υπάρχει τίποτα που να ε, υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους μηχανισμούς και, στα, και στις διαδικασίες μας. Επίσης, προτείνουμε κάποιες αλλαγές σε σχέση με την ε, δομή διακυβέρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΣΑ και γνωρίζουμε ότι εδώ στην Επιτροπή σας υπήρχαν και κάποιες προτάσεις σε σχέση με τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόταση δική μας είναι πάρα πολύ απλή. Θα εισάγουμε μια δομή διακυβέρνησης για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΣΑ που ταυτίζεται με τη δομή όλων των άλλων αποκεντρωμένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ακολουθούμε στην ουσία το μοντέλο που υπάρχει ε, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, ε, Χημικών κτλ. κτλ. Αυτή τη στιγμή ο ΕΦΣΑ είναι παρείας σε σχέση με το πώς είναι οργανωμένο το διοικητικό του συμβούλιο και πλέον ευθυγραμμίζεται το δικό του, ε, η δική του δομή οργάνωσης με εκείνη των άλλων αποκεντρωμένων οργανισμών που η δομή αυτή των άλλων οργανισμών άλλωστε έχει τύχει τη υποστήριξη της, ε, του Κοινοβουλίου. Και τέλος προτείνουμε και μια ουσιαστική αύξηση των πόρων για τον ΕΦΣΑ προκειμένου να μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντά του και αυτός ε, ξέρετε πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο χρειάζονται επενδύσεις για να ε, έχει κανείς αποτελέσματα γι' αυτό και ακριβώς επειδή θα αυξηθεί ο φόρτος εργασίας λόγω της πρότασής μας του ΕΦΣΑ, συνοδεύουμε ε, την πρότασή μας και με αύξηση ε, του κονδυλίου για τον ΕΦΣΑ. Επίσης, κοινοποίηση κινδύνων. Γνωρίζουμε ότι είναι πρόκληση των να ενημερώνει πολίτες για ε, προβλήματα ή κινδύνους που υπάρχουν στην αλυσίδα τροφίμων. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να ε, κλείνουμε τα μάτια στα προβλήματα που υπάρχουν. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα πολύ καλύτερα. Θα είναι μεγάλη πρόκληση βεβαίως να τα καταφέρουμε. Δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμα πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να αντιποκριθούμε σε ένα τέτοιο στόχο, πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε καλύτερα και με μεγαλύτερη διαφάνεια. Γνωρίζουμε όμως ότι η Κομισιόν θα χρειαστεί να προτείνει στα κράτη-μέλη και στην επιστημονική κοινότητα συγκεκριμένε προτάσει για το πώ μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Και για τον λόγο αυτό η πρότασή μας επίσης περιλαμβάνει και μια σειρά από υποπροτάσεις όσον αφορά το, το, το θέμα αυτό. Και τέλος, εκφράζουμε βεβαίως και πάλι την προσήλωσή μας στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο για τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων. Έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία μαζί σας άλλωστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα λάβουμε πλήρως υπόψη μας τις ε, ε, προτάσεις σας ε, και της δικής σας Επιτροπής και όλων των άλλων αρμόδιων, συναρμόδιων επιτροπών του Κοινοβουλίου. Και ελπίζουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας να καταφέρουμε να, να λάβουμε υπόψη μας και να εντάξουμε όλες τις προτάσεις και ιδέες που θα έχουν εκφραστεί. Ξαναλέω, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης Δεσμευόμαστε ότι θα ταξιοποιήσουμε αυτά τα περιθώρια. Είναι πολύ φιλόδοξη προθεσμία που έχουμε θέσει στον εαυτό μας, αλλά έχουμε εικόνα ότι και εσείς και το Συμβούλιο γνωρίζει τον επίγοντα χαρακτήρα αυτής της πρότασης και θέλετε κι εσείς όπως και εμείς άλλωστε να καταλήξουμε σε αποτελέσματα το δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Αν λοιπόν ο εισηγητής δεν θέλει να προσθέσει κάτι, μπορούμε να συνεχίσουμε. Όχι, ο εισηγητής. Η Κομισιόν δεν μου απάντησε σε ό,τι αφορά το ερώτημά μου για το ποιος θα χρηματοδοτήσει τις ε, μελέτες επιβεβαίωσης, την επιβεβαίωση των μελετών. Ε, και σε άλλα ζητήματα, αλλά θα συνεχίσουμε να συζητάμε αυτό το θέμα στο μέλλον, οπότε ελπίζω θα λάβω τις απαντήσεις μου. Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει τώρα για αυτό το θέμα. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, ζητώ συγγνώμη. Για το θέμα των, μελετών επιβεβαίωσης. Πράγματι, προτείναμε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλισης Τροφίμων, η ΕΦΣΑ, να διαθέτει έναν προπολογισμό για να διενεργήσει τέτοιου είδου μελέτε και γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια παράπονα σε σχέση με αυτό στην Επιτροπή σα, αλλά όχι μόνο εδώ και στην ε, Επιτροπή Γεωργία. Οπότε να σα δώσω λίγο περισσότερε λεπτομέρειε για το τι έχουμε στο μυαλό μα. Ε, δεν αμφισβητείτε το ότι είναι ευθύνη του κλάδου και του ετούντος ε, να παράσχει τα απαραίτητα επιστημονικά στοιχεία τα οποία θα ε, υποστηρίξουν το αίτημά του. Είναι προφανές ότι ο ετών θα πρέπει να αναλαμβάνει την ε, δαπάνη αυτή. Από την Ευρωπαϊκή όμως Πρωτοβουλία Πολιτών έγινε σαφές ότι μερικές φορές χρειάζονται πρόσθετες μελέτες συμπληρωματικές και βέβαια κατ' εξαίρεση δεν θα είναι αυτός ο γενικός κανόνας. Μερικές φορές μπορεί η ΕΦΣΑ, για παράδειγμα, να είναι ικανοποιημένη από τις επιστημονικές μελέτες που ε, κατέθεσε ο, ετού, ετών, παρόλα αυτά όμως να χρειάζονται πρόσθετα εχέγγυα. Εχέγγυα τα οποία θα ξεπερνούν τα δεδομένα τα οποία θα είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή. Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν υφίστανται οριζόντια ζητήματα τα οποία υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο κλάδο. Για παράδειγμα, ε, σε ουσίες ε, οι οποίες αποτελούν ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, αλλά δεν περιορίζεται η χρήση τους σε ένα μονοκλάδο και γι' αυτό το λόγο καμία εταιρεία δεν μπορεί να ε, αναλάβει το, το κόστος των ερευνών. Οι αφλατοξίνες για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι μια τέτοια ουσία. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις ίσως να χρειάζονται μελέτες επιβεβαίωσης. <clears throat> Πάντως, πρόθεση δεν είναι επουδενή να συγχρηματοδοτήσουμε τις ε, δράσεις ε, του κλάδου. Έτσι. Λυπούμαστε αν δημιουργήσαμε αυτή την λαθασμένη εντύπωση και αν μπορούμε να το διευκρινίσουμε στο κείμενο πολύ ευχαριστώ. αυτό. Σε ό,τι αφορά τη μελέτη ε, ε, ε, αντικτύπου, αναφέρθηκα σε αυτό, ίσως όχι με πολλέ λεπτομέρειες. Ε, πράγματι δεν έγινε μελέτη αντικτύπου για αυτή την πρόταση που υποβάλαμε. Γιατί είναι απάντηση στην πρωτοβουλία των πολιτών και θέλαμε η απάντηση αυτή να έρθει γρήγορα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας. Γι' αυτό λόγο δεν είχαμε αρκετό χρόνο. Όμως πρόκειται για μια πολύ στοχευμένη πρόταση και γι' αυτό το λόγο ίσως δεν είναι απαραίτητη μελέτη αντικτύπου. Για την όλη νομοθεσία περί είχαμε αυτό που ονομάζουμε fitness check, τον ε, έλεγχο καταλληλότητας, ε, ο οποίος έλεγχος οδήγησε το συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται, ότι γενικά το σύστημα λειτουργεί σωστά. Γι' αυτό το λόγο θεωρήσαμε και δεδομένη τη πίεση και του χρόνου ότι η διαβούλευση την οποία διοργανώσαμε με τους ε, φορεί φορείς, με τα κράτη-μέλη κλπ. ήταν αρκετή και δεν χρειαζόταν μελέτη αντικτύπου. Επαναλαμβάνω λοιπόν, παρόλο που δεν έχουμε τέτοια μελέτη, η διαβούλευση έγινε σε μεγάλο εύρος. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, προθεσμία για τροπολογιε 7 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι και πάλι. Κλείνουμε και το θέμα 6. Περνάμε στο σημείο 7 τη ημερησία διάταξη Σχέδιο γνωμοδότησης για την αυτόνομη οδήγηση στις ε, ευρωπαϊκές μεταφορές. Εισηγητή ο κ. Ράντεφ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε αυτό το θέμα της αυτόνομης οδηγής τον Ιούλιο, άκουσα με προσοχή όλες σας τις παρατηρήσεις. Τώρα με, το προσχέδιο γνωμοδότησης ελπίζω να έχω καλύψει τα περισσότερα ζητήματα και να έχω καταπραίνει κάπως τους φόβους σας. Πιστεύω ότι θα είδατε το τελευταίο σχέδιο και για να σας πω γιατί πρόκειται θα σας μιλήσω για τις εξελίξεις. Θεωρούμε ότι ένα επιπρόσθετο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα οδηγήσει στο να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις και κινδύνους σε σχέση με τον ε, ε, μεγαλύτερο ρυθμό αυτοματοποίησης κατά την οδήγηση. Με βάση τις ε, τεχνολογικές αλλαγές θα πρέπει να διασαφηνίσουμε ποιος θα ήταν ο υπεύθυνος ατυχήματος τη στιγμή που γίνεται ένα ατύχημα όπου συμμετέχει και ένα ε, αυτόνομο όχημα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να τροποποιηθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο και κανονιστικό πλαίσιο για να υπάρχουν νέοι κανόνες ε, περί ευθύνης, περί ευθύνης. Μία από τις λύσεις θα ήταν να εισαγάγουμε μία διευθέτηση κατά την οποία η αποζημίωση θα ορίζεται σαφώς τη στιγμή που συμμετέχει ένα αυτόνομο ε, όχημα κατά τη διάρκεια, διάρκεια ενός ατυχήματος. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει μία γενικότερη διευκρίνηση λειτουργίας των αυτόνομων οχημάτων για να μην υπάρχει κατακαιρματισμός της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα τροποποιήσουμε την ε, σύμβαση οδικών μεταφορών της ε, Βιέννης, συμπεριλαμβάνοντας και τα αυτόνομα οχήματα. Θα ήθελα να μιλήσω για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την προστασία των αυτόνομων οχημάτων έναντι των επιθέσεων στον ε, κυβερνοχώρο. Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί και μηχανήματα μάλλον καταγραφής δεδομένων έτσι ώστε να μπορέσουν να διερευνηθούν τα ατυχήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης θα πρέπει να ορίσει καλύτερα τους κανόνες προστασίας δεδομένων μέσα στα πλαίσια της αυτοματοποίησης δεδομένων και της πρόσβασης σε αυτά μέσα στα πλαίσια του κανονισμού προστασίας δεδομένων. Τέλος, όπως ισχύει και σε άλλους τομείς, θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσα στα πλαίσια της τεχνητής ευφυΐας. Όπως ξέρετε υπάρχει ένα πλαίσιο τεχνιών σε σχέση με το λογισμικό που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης. Περί αυτού πρόκειται λοιπόν και ελπίζω να είναι μια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κινηθούμε έτσι ώστε να έχουμε ένα εξαιρετικό τελικό σχέδιο γνωμοδότησης για την Επιτροπή Τραν. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέλκεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ράδευ για τη γνωμοδότησή του. Την υποστηρίζω σε γενικές γραμμές. Να υπενθυμίσω ότι ο χρόνος πιέζει. Το 2020 ε, υπάρχει στόχος να κινούνται στους δρόμους μας αυτοκίνητα αυτόματης οδήγησης ε, κατηγορίας 4. Πρέπει λοιπόν να επισφέρσουμε τις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνει η αυτόματη οδήγηση. Συμμερίζομαι την άποψη του συντάκτη ότι μια κοινή ενωσιακή προσέγγιση είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα αυτόματα οχήματα θα κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και γι' αυτό χρειάζονται και οι σχετικές τροποποιήσεις στη Συμφωνία της Βιέννης. Βεβαίως, χρειάζεται να συνοδεύεται αυτή η εναρμόνιση και από συγκεκριμένε και πολύ σαφείς ευθύνε. και ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, συμμορφωνόμαστε και με τους κανόνες για τα black box, τα μαύρα κουτιά, ώστε να μπορούν να, δια, να ε, και τα τυχόν ατυχήματα που θα συμβαίνουν. Η πρόταση της Κομισιόν άλλωστε ενέτασε αυτήν την κατηγορία και ε, σε αυτούς τους κανόνες για την ανάληψη ευθύνης. Συμφωνώ επίσης με τον ε, κύριο Ράντεφ ότι σε περίπτωση ε, πλήρους αυτόνομης οδήγησης θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιος ακριβώς θα πληρώνει τυχόν ζημίες που θα προκαλούνται. Έχω την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε μόνο στην αυτόνομη οδήγηση, χωρίς όμως να ορίζονται με σαφήνεια και οι ευθύνες που θα, που θα προκύπτουν από ε, τυχόν ατυχήματα. Και νομίζω ότι η, η ευθύνη αυτή δεν θα πρέπει να επικεντρώνεται μόνο ε, στους κατασκευαστές των, ε, των, ε, των οχημάτων αλλά θα πρέπει να αφορά και τους οδηγούς, τους κατόχους αυτών των ε, οχημάτων. Να υπενθυμίσω δε ότι το 1% των ε, ατυχημάτων μόλις ε, ευθύνεται, οφείλεται σε κακή συντήρηση ή σε τεχνικά προβλήματα. Επίσης, σημαντικό στοιχείο είναι η προστασία των θυμάτων. Γι' αυτό ε, συμφωνώ με την άποψη του κ. Ράντεφ ότι θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα συστήματα ασφάλισης. Και όπως άλλωστε έχουμε πει ω κοινοβούλιο στον τομέα της ρομποτική, θεωρώ ότι και σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, περιορισμός της ευθύνης όσον αφορά το είδος και την έκταση ε, της ζημίας που θα προκαλείται. Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, από τα δεδομένα που θα παράγει το ίδιο το όχημα, ο εισηγητής μας ε, επίσης προκρίνει μια γενική προσέγγιση με την οποία συμφωνώ, αλλά τονίζω ότι πρέπει να ελεγχθεί, να εξεταστεί αν θα μπορούσε να ε, εξασφαλιστεί και μια σύνδεση με, τον, ε, ε, με την οδηγία για τα μη προσωπικά δεδομένα. Η Επιτροπή ΙΜΚΟ μάλιστα είχε προκρίνει φέτος σε ψήφισμά της τα δικαιώματα χρήσης και όχι τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Κάτι τέτοιο, μια τέτοια ιδέα νομίζω ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτό το τομέα όσον αφορά τα δεδομένα που θα παράγουν τα ίδια τα οχήματα μέσω των αλγορίθμων τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα χρήσης θα διαμορφωθούν με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο θεμητός ανταγωνισμός, ώστε να μην δημιουργηθούν μονοπόλια και από άποψη προστασίας των καταναλωτών αλλά και από την άποψη των ανεξάρτητων συνεργείων αυτοκινήτων θα πρέπει ε, σύμφωνα και με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων να υπάρχει ελεύθερη ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά για όπως και οι κατασκευαστές θα έχουν άλλωστε τέτοια πρόσβαση και θα πρέπει ε, να εξασφαλιστεί και ε, αυτή η διάσταση προκειμένου να αποφεύγονται φαινόμενα, φαινόμενα ε, εγκλωβισμού, lock-in των καταναλωτών. Ευχαριστώ κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Ράντεφ για αυτή την γνωμοδότηση, για αυτή την έκθεσή του. Στηρίζω τα όσα είπε μόλις τώρα ο Τίμο. Συμφωνώ με, την, με το περιεχόμενο της έκθεσης. Συνεχίζει, δίνει συνέχεια στην νομοδότηση της περασμένης χρονιάς και κρίμα που δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στο, ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Γιατί από ό,τι φαίνεται πραγματικά δεν έχουμε δει πρόοδο. Ε, θέλω να προσθέσω το εξής σε ό,τι αφορά το σημείο 3 για το θέμα της ασφάλειας. Η γενίκευση των, <clears throat> ε, του τύπου ασφάλισης ε, χωρίς ε, σφάλμα ε, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Όμως ο εισηγητής λέει ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, αρκετά δεδομένα ε, για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύστημα ασφάλισης και ακόμα και αν το κάνουμε θα ήταν πολύ δαπανηρό. Ε, θα περιόριζε την πρόσβαση σε αυτά τα οχήματα μόνο σε ανθρώπους που είναι πολύ τυχαίροι και ευλογημένοι. Δεν έχω να δώσω απάντηση. Ίσως πράγματι χρειαζόμαστε μια βάση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ίσως αξίζει να το σκεφτούμε. Ευχαριστώ. Thank you as well. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Επιτροπή θα ήθελε το λόγο, ο Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για το προσχέδιο και για την συζήτηση που λαμβάνει η χώρα για το θέμα της αυτόνομης οδήγησης. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και χαίρομαι ε, ότι και εσείς και η Επιτροπή Μεταφορών το έχετε βάλει ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Θεωρούμε επίσης ότι αυτή η συζήτηση είναι η αφετηρία ενός διαλόγου που θα γίνει και για θέματα πολιτικής και για θέματα νομοθετικά καθαρά. Όπως είπατε και εσείς, ε, Έχουμε πολλά να κάνουμε σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο. Μάλιστα, θίξατε διάφορα ζητήματα. Για παράδειγμα, το καθεστώς της ευθύνη, ε, της ασφάλειας, του καταγραφέα, των οδικών κανόνων, των κανόνων κυκλοφορίας. Συμφωνούμε εν γέννη μαζί σας ε, και στην ανακοίνωση την οποία ε, δημοσιεύσαμε το Μάιο είδαμε το θέμα σε όλες του τις διαστάσεις. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ε, εμεί θεωρούμε ότι εργαζόμαστε σε τρεις παράλληλες κατευθύνσεις. Τεχνολογία και υποδομές αφενός, που είναι απόλυτα σημαντικό για να εξασφαλιστεί αυτό η Νομικό πλαίσιο ε, και τρίτον, οτιδήποτε έχει σχέση με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα που, θα, που σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε και ήδη ξεκινήσαμε από το Μάιο μέχρι του χρόνου, το Μάιο. Να σχολιάσω αυτά που είπατε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ευθύνη, νομικής ευθύνη. Η οι συνάδελφοι από την Γενική Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων μπορούν να σας πούν περισσότερα, αλλά προφανώς και εξετάσαμε διάφορε δυνατότητε ε, και σε ό,τι αφορά τα προϊόντα και σε ό,τι αφορά τα οχήματα. Και έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή αλλαγή. Αυτή τη στιγμή, τι εννοώ αυτή τη στιγμή, εννοώ το εξή: Ε, θεωρούμε ότι σταδιακά θα αυξάνονται τα αυτόματα οχήματα ε, και θα πρέπει να κάνουμε τη διάξη ανάμεσα σε αυτόματα οχήματα με οδηγό και σε αυτόματα ε, οχήματα χωρίς οδηγό. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει όταν ο οδηγός είναι απόν. Ε, για το θέμα της ευθύνη προϊόντων έχουμε ήδη δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας και εξετάζουμε το πώς θα επηρεαστεί η ασφάλεια προϊόντων από τις, από τεχνολογίες. Ε, θα περιμένουμε να δούμε τι, ποια θα είναι τα πορίσματα της ε, Επιτροπής αυτής. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των οχημάτων, συστήματα ασφάλισης οχημάτων μάλλον, ήδη υφίσταται μια δυνατότητα ε, να δοθεί αποζημίωση σε θύματα ατυχήματος ανεξαρτήτως τίτος αν μιλάμε για παραδοσιακά συμβατικά ή αυτόνομα οχήματα. Οπότε υφίσταται ένα τέτοιο σύστημα, ένα τέτοιο καθεστώς ασφάλισης. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τους καταγραφείς, απολύτως απαραίτητο για τον τομέα αυτό. Μαζί με την ανακοίνωσή μας ετοιμάσαμε και μία αναθεώρηση της γενικής νομοθεσ... κλαδικής νομοθεσίας και εκεί στην αναθεώρηση αυτή περιλαμβάνουμε και τους καταγραφείς. Θα πρέπει να δούμε όλα τα θέματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την ιδιωτικότητα και να εξασφαλίσουμε ότι ταυτόχρονα ότι ο καταγραφέας θα λειτουργεί όπως τον θέλουμε. Η Επιτροπή ΙΝΚΟ θα συζητήσει αυτό το θέμα και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τις κατεξοδότηση πράξεις. Σε ό,τι αφορά τη Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα εργασίας στη Γενέβη ε, που επεξεργάζεται κατευθυντήρες ραμές για αυτόνομα οχήματα που ενδεχομένως θα ενταχθούν στη σύμβαση. Αλλά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο επίπεδο 4, ε, στον ορίζοντα δηλαδή του 2030 και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε νομικό κείμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Το πακέτο κυβερνοασφάλειας ε, σχετικό με τα αυτόνομα οχήματα είναι κομμάτι της δουλειάς που γίνεται στη Γενέβη γιατί εκεί χρειάζονται παγκόσμια πρότυπα. Οπότε πολύ σωστά λέτε ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή προσέγγιση ώστε να μην κατακαιρματιστούμε. Θέλουμε ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την κυβερνοασφάλεια προκειμένου τα οχήματα αυτά να κυκλοφορούν ελεύθερα με τους ίδιους κανόνες. Ε, εργαζόμαστε λοιπόν επί ενός κανονισμού ο οποίος θα ε, ψηφιστεί αρχές του επόμενου χρόνου στη Γενέβη. Αυτοί είναι οι κανόνες οι οποίες θα ενταχθούν επίσης στον γενικό ε, κανονισμό του κλάδου, κλαδικό κανονισμό. Τώρα να δώσω το λόγο στην άλφα της νομικής υπηρεσίας. Δύο λόγια για την νομική ευθύνη. Μετά την έκθεση Ντελβό που υιοθετήθηκε το Φεβρουάριο, η Κομισιόν υιοθέτησε <clears throat> ένα ε, ανακοινωθέν τον Απρίλιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Το ένα τρίτο αυτής ανακοίνωση αναφέρεται σε, στο νομικό και ηθικό πλαίσιο. Η ασφάλεια και η νομική ευθύνη είναι δύο θέματα πολύ σημαντικά, δύο σημαντικές συνιστώσεις αυτού του πλαισίου. Το θέμα βέβαια είναι πολύ περίπλοκο. Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε, συστήσαμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ε, με δύο συνστώσεις. Πρώτον, ε, μία που, αφο, που ε, εξετάζει τα θέματα της ευθύνης προϊόντων και το άλλος κλάδος της ομάδας εμπειρογνωμόνων ασχολείται με πιο, μια πιο ολιστική προσέγγιση το θέμα των νομικής ευθύνης εξετάζει το κατά πόσον το συνολικό νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες και αν όχι αυτός ο κλάδος της ομάδας εμπειρογνωμόνων θα <clears throat> υποβάλει συστάσεις για το πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί το πλαίσιο και πώς θα μπορούσε η Κομισιόν να βοηθήσει σε αυτή την προσαρμογή. Μετά από δικό σας αίτημα, ε, δώσαμε πρόσβαση στο κοινοβουλικό συζητητέ και στις δύο, και στους δύο κλάδους της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Αυτοί οι παρατηρητές ήδη έχουν παρακολουθήσει τις πρώτες συνεδριάσεις ε, της ομάδας εμπειρογνωμόνων και θα σας ενημερώσουν. και για τα δύο σκέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων, τα αυτόνομα αυτοκίνητα είναι ένα παράδειγμα της δουλειά της ομάδας εμπειρογνωμόνων για να διαπιστώσουμε το κατά πόσον οι καινούργιες τεχνολογίες ε, εντάσσονται, καλύπτονται ήδη από το ισχυρό νομικό πλαίσιο. Θα συζητηθεί το θέμα των αυτόνομων οχημάτων στην επόμενη συνεδρία της ομάδας εμπειρογνωμόνων μέσα στο Σεπτέμβρη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το δούμε σε βάθος και να δούμε καταρχήν το κατά πόσον το εθνικό ή το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο επαρκεί αυτή τη στιγμή. Αν όχι, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να προσαρμοστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έκθεση Delvo και θα είμαστε ευγνώμονες και για την έκθεση την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή του κύριου Ράντεφ και περιμένουμε συνεργαστούμε στενά με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ο κύριος Λεμπρετών θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που δεν με ξεχάσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ραντέφ για την έκθεση αυτή που σχετίζεται ένα σημαντικό ζήτημα διότι αφορά τα αυτόνομα οχήματα που δεν θα αργήσουν να κυκλοφορούν στις οδικές μας αρτηρίες ε, και θα ήθελα να πω ότι το δίκαιο δεν έχει προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά την αστική ευθύνη. Εκτιμώ το γεγονός ότι ο κύριος Ραντεφ μιλά για ένα, θέμα, για ένα ζήτημα υποχρεωτικής ασφάλισης. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Θα ήθελα όμως να κάνω ε, ορισμένα σχόλια για τις τρεις μου τροπολογίες. Εάν θέλουμε να διασαφηνίσουμε το θέμα της αστικής ευθύνης και να υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση, θα αφορά την αποζημίωση των θυμάτων. Και δυστυχώς η λέξη θύμα δεν υπάρχει στο σχέδιο γνωμοδότησης, διότι αυτό είναι το τελικό μας μέλημα, να μας απασχολήσει η τύχη των θυμάτων. Επίσης, όταν μιλάμε για απόδοση ευθυνών, θα πρέπει να ξέρουμε πώς θα γίνει αυτή η απόδοση. Γιατί μπορεί να ισχύσει η λογοδοσία για τον ιδιοκτήτη, το χρήστη ή τον κατασκευαστή των οχημάτων αυτών. Θα πρέπει να ξέρουμε πού θα αποδώσουμε την ευθύνη ή πώς θα την κατανείμουμε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχει και ένα άλλο έλλειμμα, μία έλλειψη μάλλον, δηλαδή το θέμα του νομικού προσώπου πίσω από κάθε αυτόνομο όχημα. Ορισμένα ε, λόμπι δεν θέλουν ο άνθρωπος να φέρει ευθύνη και θα ήθελα να πω ότι το, σύμφωνα με το γαλλικό δίκαιο ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της αστικής ευθύνης δεν αφορά μόνο την αποζημίωση αλλά και τις κυρώσεις, ένα κυρωτικό πλαίσιο, δηλαδή να ορίζει τους υπευθύνους και κατά την άποψή μου την ευθύνη δεν μπορεί να φέρει παρά άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να σας ξαναπώ ότι η προθεσμία τροπολογιών είναι η 6η Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ και συνεχίζουμε με το θέμα υπάρχει μόνο 8 τροπολογίες σε σχέση με διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Χρυσόγονος είναι ο εισηγητής, ο οποίος δεν είναι παρόν. Ο κύριος Μαστάλκα τον αντικαθιστά. Ωραία. Komluvil kolegu který tu dnes námi nemůže být. Ε, Πράγματι εκπροσωπώ τον κύριο Χρυσόγωνο. Δυστυχώς ε, δεν μπορεί να παραστεί. Σήμερα μου ζήτησε να διαβάσω τα σχόλια του στα αγγλικά. Ίσως ήθελε να με, να με τιμωρήσει. Ε, οπότε, θα ήθελα να, λέω και ο Σόνς, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Θα προσπαθήσω να τις λάβω υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Ε, στις συμβαστικές προτάσεις θα υποβάλλω. Ο βασικός ε, στόχος είναι να βελτιωθούν αποτελεσματικά οι προτάσεις Κομισιόν για μια οδηγία για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα στηρίξω την τροπολογία, τις τροπολογίες που προωθούν πιο διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας και προσφέρουν επαρκή προστασία σε όλους τους εργαζόμενους. Η παραγωγικότητα, ε, η μακροχρόνια παραγωγικότητα ε, εμπλέκει και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προασπιστεί ε, περισσότερο αν συνδυαστεί με την αποτελεσματική εφαρμογή του χάρτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εργάζεται με συνθήκε που θα σέβονται την αξιοπρέπειά του, την ασφάλειά του και την υγεία του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you as well. Uh, Thank you very much. Um, I would like to start with... ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεση αυτή. Είναι πολύ καλή. Όμως Στη Σουηδία έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο αγοράς εργασίας και για μας είναι απαραίτητο η οδηγία αυτή να σέβεται το δικό μας μοντέλο που εμπεριέχει και περιλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους, το δικαίωμά τους να εισέρχονται σε διαπραγματεύσεις και να ε, συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν πλήρες δικαίωμα να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο κατάλληλο επίπεδο και θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν τη δυνατότητα να ε, ικανοποιούν τις απαιτήσεις, τις απαιτήσεις αυτής της οδηγίας και να, να προστατευτούν τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών. Να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων, της προστασίας συμφερόντων των εργαζομένων και των εργοδοτών. Και σε αυτό το πλαίσιο έχω υποβάλει κάποιες ε, τροπολογίες, την 115, την 134 και την 226. Και θα ήθελα να σας καλέσω να τις υπερψηφίσετε, γιατί για εμάς στη Σουηδία ε, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δεν καταλαβαίνω ε, σε ποιον ακριβώς τομέα των αρμοδιοτήτων της Γιούρη εμπίπτει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά ίσως δεν καταλαβαίνω πολύ καλά την ε, διάκριση αυτών των αρμοδιοτήτων μεταξύ των Επιτροπών του Κοινοβουλίου. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή μέσω του εκπροσώπου του και όλου όσου έχουν υποβάλει τροπολογίε τι οποίε και διαβάσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Κάποιε παρατηρήσει διευκρινιστικού χαρακτήρα. Πρώτον, κάτι που συνδέεται με το τελευταίο σας σχόλιο. Βρισκόμαστε πλέον στον τομέα των ε, όρων εργασίας. Και εδώ η αρμοδιότητα προβλέπει μόνο ελάχιστες απαιτήσεις, ελάχιστα πρότυπα. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν προτείναμε να ευθυγραμμίσουμε την πρότασή μας με αυτό το γεγονός και να ενισχύσουμε στην ουσία τη θέση των εργαζομένων, σε εκείνων που εργάζονται σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αλλά δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να προτείνει μόνο ελάχιστα ε, πρότυπα. Βεβαίως από εκεί και πέρα υπάρχουν μεγάλα ε, περιθώρια προσαρμογής και ευελιξίας για τα κράτη-μέλη. Και με αυτό περνάω στη δεύτερη παρατήρηση, στην οποία θέλω να σταθώ, που σχετίζεται με τους κοινούς κοινωνικούς εταίρους. Βεβαίω, ο κοινωνικό διάλογο εξακολουθεί να μα ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραβιαστούν ε, τα διάφορα μοντέλα αγοράς εργασίας που υπάρχουν. Και γι' αυτό το λόγο η οδηγία μας, η οδηγία που προτείνουμε, προβλέπει το χώρο για την προσαρμογή των προτύπων αυτών ε, μέσω συλλογικών ε, συμβάσεων. Και στο Συμβούλιο τα περισσότερα κράτη-μέλη μας έχουν δηλώσει ότι αρκεί μια τέτοια πρόβληψη. Καταλαβαίνω ότι δεν, δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πάντες, αλλά αν μια χώρα όπως η Δανία που έχει τους κοινωνικούς εταίρους στο επίκεντρο της νομοθεσίας της μπορεί να υποστηρίξει αυτή την πρόταση ε, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι ισορροπημένη η πρότασή μας φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε τυχόν βελτιώσεις που θα μπορούσαν να, να ενισχύσουν την ε, πρόταση δεδομένου όμως πάντοτε ότι πρόκειται για ενωσιακή νομοθεσία και νομοθετούμε και για εργαζόμενους που εργάζονται σε κλάδους ε, όπου δεν υπάρχει εναρμόνιση. Θέλουμε να προστατεύσουμε και αυτούς. Ε, σταματώ εδώ. Αν βεβαίως ε, θέλετε περαιτέρω διευκρινήσεις, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Να πω ότι η έγκριση στην Επιτροπή Γιούρι προβλέπεται να γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου. Και συνεχίζουμε με το σημείο 9. Εξέταση σχεδίου έκθεσης για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στο εταιρικό δίκαιο. Η είναι ο κύριος Σβιέφκα. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη μου χαρά θα σας παρουσιάσω τα σχόλιά μου σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το εταιρικό δίκαιο. Στόχοι είναι οι εξής. Προβλέπονται διάφορες διευκολύνσεις τις οποίες περιμένουν οι επιχειρήσεις μας. Υπάρχουν, υπάρχει μια σειρά από εργαλεία τα οποία μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Η πρόταση αυτή συμβάλλει στην ενίσχυση ε, της ενιαίας αγοράς. Αυτές είναι, αυτή είναι η στόχη, λοιπόν. Τα σημαντικότερα ζητήματα είναι τα εξής. Πρώτον, μιλάμε για την online εγγραφή, καταχώρηση ε, μιας εταιρείας και των υποκαταστημάτων της. Άλλο σημαντικό στοιχείο σχετίζεται με την αρχή άπαξ που εισάγεται για πρώτη φορά εδώ. Βάσει αυτής της αρχής Μάλλον, ο μη σεβασμός αυτής της αρχής πολλές φορές ε, αυξάνει τη γραφειοκρατία, την διοικητική επιβάρυνση, γιατί ακριβώς χρειάζεται κανείς να επαναλαμβάνει τις ίδιες διαδικασίες πολλές φορές. Το έγγραφο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάρα πολύ καλό. είναι ένα έγγραφο υψηλής ποιότητας. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να πω ότι εμείς στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουμε ως στόχο να αποσαφηνίσουμε κάποιες διατάξεις, ώστε αυτές να είναι πρακτικά εφαρμόσιμες. Θα πρέπει να είναι πέρα για πέρα σαφές, επίσης, ποιες ακριβώς θα είναι οι υποχρεώσεις των εμπλεκομένων. Αυτό βεβαίως αφορά κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των επιχειρηματιών της Ευρώπης. Το έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Η Κομισιόν άλλωστε έχει διεξαγάγει και μελέτες σε σχέση με αυτό το θέμα και διαβουλευσει. Ο γενικός σκοπός είναι να εξασφαλίσουμε την νομική συμβατότητα βεβαίως αλλά και την συνεκτικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου και τη συμβατότητα μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Για να μπορέσει το σύστημα αυτό της online καταχώρησης να λειτουργήσει, χρειαζόμαστε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες, κάποια εχέγγυα. Να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που θα, παρέχονται και θα υποβάλλονται θα είναι ακριβείς. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση να υπάρχουν κίνδυνοι. Θα πρέπει όλοι να μπορούν να είναι βέβαιοι ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Μητρό είναι σωστές και ακριβείς. Έχω υποβάλει και κάποιες τροπολογίες με σκοπό ακριβώς να αποσαφηνίσουμε κάποιες από τις διατάξεις. Ιδίως όσον αφορά τα υποκαταστήματα. Τα είχα πει και πριν τις θερινές διακοπές. Οι διατάξεις που αφορούν τα υποκαταστήματα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφής. Όσον αφορά την υποβολή εγγράφων τεκμηρίωσης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντοτε η αυθεντικότητα και η ακρίβεια του φακέλου που υποβάλλεται. Η γνησιότητα, η ακρίβεια και η αυθεντικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα τρία στοιχεία και γι' αυτό και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση. Όλες οι διαδικασίες επίσης θα πρέπει να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία. Αλλά θα πρέπει να συμμορφώνεται και με τον κανονισμό για την ε, ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Σκοπός μας λοιπόν είναι να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ διαφορετικών φορέων. Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και στις επιχειρήσεις μας. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με μια οδηγία, με μια πρόταση οδηγίας. Τα ηχέγγυα που προβλέπονται σε αυτήν θα λειτουργήσουν μόνο αν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Οι απαιτήσει λοιπόν που ανέφερα και νωρίτερα πιστεύω ότι θα πρέπει να βασίζονται στην εθνική νομοθεσία και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Πολλά κράτη-μέλη διαθέτουν πολύ σαφείς διατάξεις και κανόνες για την online καταχώρηση. Κάποια κράτη-μέλη δεν διαθέτουν ακόμη. Θα χρειαστεί να τους θεσπίσουν αυτούς τους ε, κανόνες κατά τη μεταφορά της συγκεκριμένη οδηγίας στο εθνικό του δίκαιο. Γεγονός είναι ότι οι επιχειρήσεις μας χρειάζονται ασφάλεια δικαίου και χρειάζεται να γνωρίζουν ποιες ακριβώς είναι οι υποχρεώσεις τους. για την απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Όταν ένα κράτος μέλος ρωτά κάποιο άλλο κράτος μέλος αν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο έχει στερηθεί του δικαιώματός τους να, ασκηθεί, να ασκεί συγκεκριμένο επάγγελμα. Αν η απάντηση είναι θετική, θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη σχετική αιτιολόγηση. Για ποιο λόγο έχει ε, αφαιρεθεί το δικαίωμα άσκηση ενό επαγγέλματο από κάποιο πρόσωπο. Και στη βάση ποιων κανόνων νομικών. Εδώ υπάρχουν αποκλίνουσες ε, διατάξεις και κανόνες ε, σε επίπεδο κρατών μελών. οι λόγοι για τους οποίους μπορεί κανείς να στερεθεί του δικαιώματο του να ασκεί επάγγελμα μπορεί να διαφέρουν και να ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να προσθεθεί στην πρόταση της Κομισιόν ένα επεξηγηματικό σημείωμα. Επίσης θέλω να σταθώ σε ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα. οι απαιτήσει που σχετίζονται με την ε, υποβολή λεπτομερών αιτήσεων ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο Μητρό. Εκεί υπάρχει ένας κατάλογος ε, εγγράφων που θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν. δωρεάν. Νομίζω ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να διευρυνθεί και έχω υποβάλει και σχετική τροπολογία. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο για μια διαδικασία αφαιρεγγιότητας θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να είναι δωρεάν διαθέσιμο. Κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, κάποιοι συνάδελφοι μάλλον, θα ήθελαν να γίνουν ε, δωρεάν διαθέσιμα και άλλα έγγραφα, όπως για παράδειγμα το καθεστώς εργασίας. Αυτό νομίζω ότι υπερβαίνει τα όρια, θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρή μια τέτοια διαδικασία και επίσης οι, οι πληροφορίες αυτές ε, αλλάζουν ε, πολύ γρήγορα. Όπως και να έχει, ακούστηκαν από τους συναδέλφους πάρα πολλά σχόλια Περιμένω να ακούσουμε και πολλά ακόμα σχόλια, τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα εμπλουτίσουν το έργο μας και το κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε. Να τονίσω επίσης ότι πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η εφαρμογή και οι σχετικές προθεσμίες που έχουν τεθεί. Υπήρξε ε, πρόταση να ε, εφαρμοστεί η οδηγία αυτή σταδιακά. Κατά τη γνώμη μου όμως η οδηγία αυτή θα πρέπει να ε, εφαρμοστεί ε, στο σύνολό της. Αν χρειάζεται μπορούμε να παρατείνουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύω. Αλλά όταν γίνει αυτό θα πρέπει όλη η οδηγία να ε, τεθεί σε ισχύ. Τροπολογίες μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιούτελαντ. First of all, uh, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Σβιέφκα, για αυτή την πολύ καλή έκθεση. Υπάρχουν ε, αρκετά θετικά στοιχεία στην έκθεση, τα οποία υποστηρίζω ε, στην τροπολογία 2 σε σχέση με την δυνατότητα εναλλακτικών μέσων ταυτοποίησης, ως δηλαδή το σκανάρισμα των διαβατηρίων για παράδειγμα. Χαίρομαι για αυτή τη διαγραφή. Επίσης, άλλα μέσα ταυτοποίησης, εάν ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τότε ίσως θα μπορούσαν να εγγραφούν εταιρείε στο έδαφος τους με μειωμένες προαπαιτήσεις. Δεν θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε κίνητρα για έναν αγώνα προς τα κάτω ως προς τις προαπαιτήσεις. Θα πρέπει να γίνει ένας αγώνας προς τα πάνω. Σας ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη διαγραφή. Με απασχολεί επίσης, με απασχολούν τομείς όπου δεν συμφωνούμε. Για παράδειγμα, η τροπολογία 18 είναι πολύ προβληματική γιατί διαγράφει την αναφορά στο άρθρο 19 ε, παράγραφος 2 σημείο G σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων. Με βάση την διαφάνεια που θα πρέπει να υπάρχει ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα μέσα στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης, θεωρώ ότι οι πληροφορίες που αφορούν ε, τα μητρό εγγραφής θα πρέπει να επεκταθούν και στα, στις ετήσιες εκθέσεις, πληροφορίες για τους εργαζόμενους, καθώς και διαβουλεύσεις για τις ενδεχόμενες συμμετοχές. Άρα δεν βρισκόμαστε στο ίδιο επίπεδο. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξαιρέσουν ορισμένους τομείς όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος για απάτες με τη δημιουργία επιχειρήσεων. Μόνο τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να, να έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να ορίσουμε την έδρα και να ελέγξουμε την εταιρική βάση. Θεωρώ λοιπόν ότι αν ε, αρχίσουμε να διευρύνουμε εδώ, ίσως θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα με απάτες. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε με φυσικά πρόσωπα, κάτι δηλαδή επί του οποίου υπάρχει έλεγχος και θα δούμε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την έκθεση καθώς και, για, ε, και ως προς την ε, ανακοίνωση της προθεσμίας υποβολής τροπολογιών. Ε, ο κύριος Ράντεφ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Ταντέους για αυτή την εξαιρετική έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Θα ήθελα να πω ότι η έλλειψη κανόνων σε σχέση με την online εγγραφή καθώς και την αποκάλυψη εγγράφων οδηγούσε σε μια μεγάλη, με ένα μεγάλο κατακαιρματισμό στα κράτη-μέλη και υπήρχαν και επιπρόσθετα βάρη και δαπάνες, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που ήθελαν να διευρύνουν τις δραστηριότητες τους μέσω θυγατρικών. Αυτό ίσως οδηγήσει σε ε, ε, αποφυγή επιχειρηματικών δυνατοτήτων τη στιγμή που ορισμένες εταιρείες δεν μπορούν να εγγραφούν καν. Πολλές χώρες, αρκετές χώρες έχουν εισαγάγει τη διαδικασία επιγραμμικής εγγραφής, όπως η Βουλγαρία, η χώρα μου. Η υποβολή αιτήσεων είναι μία πιο δαπανηρή διαδικασία όταν γίνεται επί χάρτου και οι επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ε, κάνουν εγγραφή online καταβάλουν, μάλλον έχουν περισσότερα έξοδα. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία προθεσμία των πέντε εργασίμων ημερών έτσι ώστε οι ΜΜΕ να είναι πιο ανταγωνιστικές. Όμως η εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων θα πρέπει να συνοδεύεται από προστασία από κατάχρηση και απάτες. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες χωρίς χρηματική επιβάρυνση. Σε σχέση με την online εγγραφή και για τις ε, θηγατρικές εδώ μπορούμε να έχουμε να κάνουμε με οντότητες που μπορούν να εγγραφούν ανεξάρτητα από την ε, νομική τους, ε, νομική τους σύσταση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι και εγώ καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την έκθεση. Είναι εξαιρετική. Ίσως υποβάλλω κάποια τροπολογία. Δύο θέματα είναι αυτά που με απασχολούν συγκεκριμένα και συμφωνώ με τον συνάδελφο Ράντεβ, η ταυτοποίηση είναι κρίσιμο ζήτημα, δηλαδή η αξιοπιστία της ε, γνησιότητας των εγγράφων θα πρέπει να εξασφαλίζεται και στις διαδικασίες ε, online καταχώρησης εγγραφής και θα πρέπει να διακρίνεται ε, να, να, να γίνεται και μια διάκριση ανάμεσα στην έναρξη των εργασιών μιας επιχείρησης και τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της και πιστεύω ότι σε κάποιες περιπτώσεις όταν υπάρχουν αμφιβολίες θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να ζητούν και εντύπωση τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό για λόγους ασφάλειας δικαίου, εμπιστοσύνης απέναντι σε αυτά, αυτές, σε αυτά τα δημόσια μήτρο. Και βεβαίως σε πολλές χώρες ε, σημαντική, διαδικασία, σημαντική συμμετοχή στη διαδικασία μάλλον έχουν και οι συμβολιογράφοι. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό τα κρατημέλη να έχουν τη δυνατότητα να εμπλέκουν στη διαδικασία αυτή και τους συμβολιογράφους. Ε, και στην αιτιολογική έκθεση θα ήταν καλό να αναφέρεται αυτό και στα, στο διατακτικό ε, της οδηγίας. Συνολικά όμως ε, βεβαίως έχουμε να κάνουμε μια πολύ καλή έκθεση. Και σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε την εμπιστοσύνη στα δημόσια αυτά μητρώα που θα τηρούνται μέσω της αξιοπιστίας των δεδομένων που θα περιλαμβάνονται σε αυτά, την, τη γνησιότητα των εγγράφων που θα υποβάλλονται και νομίζω ότι αν τα καταφέρουμε θα έχουμε ε, ωφελήσει σημαντικότατα την ενιαία αγορά. Ευχαριστώ. Κομισιόν, θέλετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για αυτή την έκθεση και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας για τα σχόλιά τους να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Καταρχήν, ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις τις οποίες ε, προτείνει ο εισηγητής, ε, σωστά τις εντοπίζει, θα τις εξετάσουμε. Αναφέρεται όμως και στην ημερομηνία εφαρμογή. Να σας εξηγήσω το εξής. Εμείς προτείνουμε μια προοδευτική εφαρμογή, διότι γνωρίζουμε πως ένα τμήμα των μέτρων είναι πιο περίπλοκο και πιο δαπανηρό για τα κράτη-μέλη εξαιτίας του ότι χρειάζονται μηχανές ανάγνωσης κλπ. Θα δούμε τι θα πει και το Συμβούλιο. Δύο θέματα τώρα τα οποία εθίγησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Πρώτον, για αυτό που ο κ. θα διαπιστώσατε ότι στην πρόταση δεν σκεφτήκαμε καν να περιορίσουμε τις προτάσεις μας στα φυσικά πρόσωπα και να εξαιρέσουμε τα νομικά πλαίσια. Γιατί, γιατί έτσι όπως το βλέπουμε εμείς, η πρόταση θέλει να κάνει διαθέσιμα τα ψηφιακά εργαλεία και να μεταφέρει τις διαδικασίες σε ένα ψηφιακό περιβάλλον. Αν λοιπόν προκύψουν κάποια πρόσθετα προβλήματα με συγκεκριμένους τύπους εγγραφής, τότε θα πρέπει αυτά να ρυθμιστούν μέσω της πρότασης με τη χρήση και πάλι ψηφιακών εργαλείων, αλλά με προσπάθειες να λυθούν αυτές οι πρόσθετες επιπλοκές. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πώς είναι δυνατόν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν με τη χρήση των ίδιων ψηφιακών εργαλείων. Θα το φροντίσουμε, όπως σας λέω. Και μετά ένα άλλο σχόλιο, στο οποίο αναφέρθηκε η κυρία Νίμπλερ, για τους μηχανισμούς ελέγχους σε εθνικό επίπεδο. Όταν επεξεργαζόμασταν την πρόταση, προσπαθήσαμε να δούμε πώς τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή ελέγχουν τη φερεγγιότητα ή την αξιοπιστία των εγγράφων τι είδου ελέγχους διαθέτουν. Γιατί υπάρχουν τέτοιου είδου μηχανισμοί, έτσι, σε κράτη-μέλη. Και τους λάβαμε υπόψη στην πρότασή μα γιατί στόχο μα είναι πραγματικά τα εργαλεία <clears throat> να γίνουν πιο εύχριστα για τις επιχειρήσεις, αλλά να επαφίεται στα κράτη-μέλη και, και η δυνατότητα να διοργανώσουν τον έλεγχο με τον, κατάλληλο, τον πιο κατάλληλο τρόπο. Αν θέλετε να το διευκρινίσουμε βέβαια αυτό, στην πρόταση πολύ ευχαριστώ. Thank you Πρόεδρος, όπως είπε ο κ. Ζιεύκα, προθεσμία για τις τροπολογίες σας 11 Σεπτεμβρίου. Κ. Ζιεύκα, θέλετε το λόγο, ναι. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια των συναδέλφων. Εστίασαν σε θέματα τα οποία μας αποσχολούν εξ αρχής. Η αναφορά στην εθνική νομοθεσία είναι πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα την αυθεντικότητα των εγγράφων και των πληροφοριών που προσφέρονται. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιγραμμικής εγγραφής, επίσης είναι δυνατόν να ζητηθεί από το σύστημα, από τον τόντα, να υποβάλει και σε χαρτί τα έγγραφα τα οποία υποβάλλει ηλεκτρονικά καταρχήν όταν υπάρχουν κάποιες υποψίες ή για διάφορους άλλους λόγους. Ιδιαίτερος αν αυτό το άτομο δεν πληρεί τις προϋποθέσεις του εθνικού νόμου. Υπάρχουν μηχανισμοί ασφάλειας που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να κάνουν τους κατάλληλους ενέχους. Όταν δούμε τις τροπολογίες σας θα ξαναδούμε την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος περνάμε στη σημείο 10. Έκθεση για τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Κυρία Ρέγνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επάνωδο στους συναδέλφους. Έχουμε το πακέτο για το εταιρικό δίκαιο θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να επιταχύνουμε τώρα που έχουμε τα νομοθετικά κείμενα μπροστά μας. Η κατάσταση για τις εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και είναι μέχρι τώρα ε, δύσκολη όταν μια εταιρεία προσπαθεί να μεταφέρει τις δραστηριότητε της διασυνοριακά εντός της ενίας αγοράς. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου ευρωπαϊκή. Δηλαδή οι εταιρείε θα πρέπει να αλλάξουν νομική μορφή. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά. Τι χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο που θα επιτρέψει εταιρείε να μετακινούνται διασυνοριακά. Αυτό το κείμενο έλειπε και το έχουμε μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Ας δούμε λίγο το ιστορικό. Η ανάγκη πλευράς αγοράς είναι σαφής ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ούτε το Συμβούλιο ε, ε, ε ήταν τα όργανα που ξεκίνησαν αυτή τη διαδικασία. Ήταν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο με την ε, νομολογία του πυροδότησε την υποβολή αυτών των προτάσεων. Και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν υπέβαλε την ε, πρότασή της προκειμένου δηλαδή να διευκρινίσει την κατάσταση κατόπιν αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εμείς ως νομοθέτης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η ρόλη θα είναι σαφής θα επιτρέπουν αφενός τις εταιρείε να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης εγκατάστασης, δεύτερον να διευκολύνουν και να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για τις εταιρείε και τα κράτη-μέλη και τρίτον να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τους πιστωτές και τους ε, ε μετόχους μειοψηφίας των εταιριών. Η έκθεση είναι μακροσκελής, ε, δεν μπορώ να τη σχολιάσω όλη βέβαια, γιατί πρέπει να καλύψουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν θα πρέπει να ενισχύσουμε τη διαβούλευση και την ενημέρωση με, τον, ε, με τους εργαζόμενους. Με αυτές τις τροπολογίες θέλω να προστατεύσω τα συμφέροντά τους έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εκπροσώπησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο τη εταιρεία. Ήδη υπάρχει σε 7 κράτη-μέλη. Αυτό που συμβαίνει και με την ψηφιοποίηση, όπου 17 κράτη-μέλη ήδη έχει γίνει δουλειά, έτσι έχουμε και εδώ 17 ε, κράτη-μέλη έχουν ήδη νομοθετήσει, όχι 7, 17 κράτη-μέλη έχουν ήδη νομοθετήσει την παρουσία των εργαζομένων στα διοικητικά συμβουλία. Δεύτερον, θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για την ε, μετατροπή συγχώνευση ή διάσπαση εταιριών Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια παρόμοια δικασία για όλες τις ε, μεταφορές καταστατικής έδρας που θα περιλαμβάνει την, το ίδιο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων εργαζομένων. Όχι λοιπόν ε, ένας, ε, μια κούρσα προς τα κάτω, αλλά μια κούρσα προς τα πάνω. κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητάει περισσότερες πληροφορίες και να δια... ζητά τη γνώμη εκ... Ε, εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι απαραίτητο αυτό, δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά ε, είναι ε, δυνατό. Θα συζητηθεί πολύ το θέμα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, αλλά το δικό μου συμπέρασμα είναι αυτό ακριβώς. Θέλουμε επίσης να αποφύγουμε τις εταιρείες, ε, εικονικές εταιρείες. Για να αποφύγουμε τις εικονικές εταιρείες, εισάγω μια απέτηση πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας ε, στην ε, χώρα στην οποία εγγράφεται η εταιρεία. Cadbury Schweppes ήταν η, η υπόθεση στην οποία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανέφερε πως η ελευθερία ε, καταστατικής έδρας εγκατάστασης προαπαιτεί ε, την ύπαρξη οικονομικών δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη χώρα. Η οδηγία θέλει να αποφύγει το φαινόμενο Delaware, δηλαδή οι εταιρείε να εξετάζουν πού, τους βολεύει, βολεύει περισσότερο, να έχουν την καταστατική τους έδρα, που η νομοθεσία είναι λίγο πιο ευνοϊκή σε ό,τι αφορά την κοινωνική ασφάλιση, τα δικαιώματα των κλπ. κλπ. Γι' αυτό άλλωστε υποβλήθηκε και το πακέτο αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών να προσελκύσουν εταιρείε χαμηλώντα τον πύχη. Εταιρείε ε, νομικών συμβουλών, δικηγόρων κλπ. ιδιαίτερα προσπαθούν να βρουν το πιο ευνοϊκό καθεστώ. Σε ό,τι αφορά τι διασπάσει δεν βλέπω καμία προσθέμενη αξία, οπότε η πρόταση δεν αφορά τι διασυνορικές ε, διασπάσεις και προτείνω να διαγραφούν από το κείμενο. Τέλος, πολλές τροπολογίες αφορούν την διευκρίνηση των όρων και των ορισμών. Τίποτα το ιδιαίτερα πρωτότυπο, αλλά είναι τόσο σημαντικό αυτό το πακέτο που θα πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, πολύ κατανοητοί. Γι' αυτό το λόγο προτείνω συγκεκριμένες διευκρινήσεις. Στο άρθρο 2. Προστασία των άλλων ενδιαφερομένων μερών, εμπλεκομένων μερών, είναι πολύ σημαντική. Ε, πιστωτές ε, και μέτοχοι το Ε, θα πρέπει να έχουν δικαιώματα εξόδου και πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους. Ε, σας μιλώ αγγλικά σήμερα, γιατί, γιατί εργαζόμαστε στα αγγλικά ε, και είναι πιο πρακτικό να συνεχίσουμε έτσι. Αυτές είναι οι προτάσεις μου. Η, το πρωτότυπο κείμενο της έκθεσης είναι το αγγλικό, θα συνεχίσουμε έτσι. Σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίε, νομίζω ότι στην έκθεση ανέφερα άλλη ημερομηνία, αλλά νομίζω ότι η σωστή ημερομηνία ε, είναι ψηφοφορία να γίνει το Νοέμβρη, νομίζω 20 Νοεμβρίου αν θυμάμαι καλά, Τρίτη, τη δεύτερη μέρα. Και νομίζω Προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 14 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους και ηγητέ. Ε, μιλώ εδώ και πολλή ώρα, μακρηγορώ, διότι πράγματι η έκθεση είναι μεγάλη, η πρόταση είναι σημαντική και είναι σημαντικό να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας μας. Ε, thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ μας άρεσε το ότι μιλήσατε στα αγγλικά. Κύριε Ντεγκράντες, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν θα μιλήσω... Αγγλικά θα μιλήσω στη γλώσσα του Θερβάντες, γιατί έτσι θα μπορέσουν να δουλέψουν και οι διερμηνείς μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ρέγνερ για την εργασία της. Ε, θα ήθελα να πω ότι ε, προσπαθήσαμε να επιλύσουμε ζητήματα τα οποία είχαν βρεθεί εν κενό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω ότι μετά από τις συζητήσεις με την Κομισιόν είδαμε ότι θα πρέπει να υποβάλουμε δύο διαφορετικά σχέδια και όχι ένα πακέτο. Πρόκειται για ζητήματα τα οποία είναι πολυσχηδή, όπως ε, φαίνεται και από την έκθεση του κυρίου Σβιεύκα, γιατί η Επιτροπή μας έδωσε μία ξεχωριστή ε, διατύπωση σε σχέση με τα δύο αυτά σχέδια. Θεωρώ ότι η οδηγία αυτή είναι ευρύτατη και πιο ευρεία από, από την εργασία που έκανε η εισηγήτρια. Έχουμε πληθώρα ρογιών σε σχέση με και με το θέμα της νομιμότητας και του θεμητού των εργαζομένων, του θεμητού της παρέμβασης των εργαζομένων. Υπάρχουν όμως ορισμένα ζητήματα που με απασχόλησαν ως κοιόδη και ε, στην ομάδα μας θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιπρόσθετοι περιορισμοί που περιστέλουν ε, τα ευεργετήματα τα οποία αρχικά είχε προβλέψει η Επιτροπή. Θα προσπαθήσω λοιπόν, Πρόεδρε, να ε, προβάλλω αυτά τα ζητήματα εμπεριστατωμένα. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν εναρμονισμένοι κανόνες για τις διασπάσεις στα πλαίσια των διασυνοριακών συναλλαγών, έτσι ώστε να υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία των εταιριών στα πλαίσια και των διασυνοριακών μεταφορών. Σε σχέση, σε σχέση τώρα με τις ε, διασυνοριακές διασπάσεις, θεωρούμε ότι θα πρέπει να μπορούν να γίνουν μετατροπές τη στιγμή που μεταφέρεται η έδρα από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο. Θεωρούμε ότι η τελευταία ε, ερμηνεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Hollywood ήταν πολύ καλή. Επίσης, το ΔΕΚ υπερασπίστηκε την αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης για να καταπολεμηθεί η απάτη. Επίσης, θεωρούμε ότι τεχνητές λύσεις δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σε σχέση τώρα με τις διοικητικές ρυθμίσεις ως προς τις μετατροπές και τις μεταφορές, δεν βλέπουμε γιατί θα πρέπει να υπάρχουν δύο ξεχωριστές εκθέσεις. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μία έκθεση και για τους μετόχους και για τους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να υπάρχει ε, η γνώμη των αρμοδίων αρχών κατά περίπτωση και αυτό αφορά και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμενες που θα μπορούν να δράσουν αυτόνομα για να μπορέσουν να οριστούν επαρκώς επιμέρους ζητήματα. Τώρα, για να μπορούν οι μέτοχοι να βγουν από οποιοδήποτε σχήμα, θεωρούμε ότι αυτό το θέμα είναι ύψης της σημασίας για να μην διακυβευτεί το όλο εγχείρημα. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ συμφερόντων των ε, μετόχων που θέλουν να αποχωρήσουν και των μετόχων που θα πρέπει να παραμείνουν. Επίσης, οι πιστωτές θα πρέπει να τύχουν προστασίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσφύγουν σε δαπανηρά μέτρα. Οι πιστωτές θα πρέπει να έχουν την ίδια δύναμη με τη δύναμη της αρχικής αξίωσης. Τέλος, θεωρώ, κυρία εισηγήτρια, ότι είναι πολύ καλή εργασία σας, είναι συμπληρωματική ε, σε σχέση με την εργασία της Κομισιόν, αλλά κυρία Ρέγνερ μπορείτε να βασιστείτε και σε εμάς για να φτάσουμε σε μια συμφωνία σε σχέση με την κινητικότητα και την επιχειρηματική λειτουργικότητα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια καλύτερη λειτουργία της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, κάτι το οποίο και εμείς υποστηρίζουμε όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Η Επιτροπή θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ ιδιαίτερα και την εισηγήτρια για αυτό το ζήτημα και την ε, σκόπιμη ανταλλαγή απόψεων με όλους τους συνομιλούντες. Όπως ε, μιλήσαμε και, στην, ε, για την προγενέστερη έκθεση, οι δύο αυτές εκθέσεις αποτελούν πακέτο που προέβαλε η Επιτροπή και χαιρόμαστε γιατί και οι δύο ε, εισηγητές είναι φιλόδοξοι και θέλουν να προχωρήσουμε γοργά. Αυτά είναι ζήτημα τα οποία έχουμε συζητήσει επί μακρόν. Η Επιτροπή έχει προβάλει διάφορα σχήματα σε σχέση με το εταιρικό δίκαιο και χαιρόμαστε γιατί και η Επιτροπή σας είναι πολύ φιλόδοξη. Τώρα, σε σχέση με το σχέδιο γνωμοδότηση, σε σχέση με τις μετατροπές συγχωνεύσεις και διασπάσεις, χαιρόμαστε γιατί η εισηγήτρια αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία της πρότασής μας, γιατί πρόκειται και για δύο εκκλήσεις που είχαν γίνει από εσάς, τις οποίες αναγνωρίσαμε. Πρόκειται για μία περίπλοκη έκθεση. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, απλώς να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν θα ήθελα να πω, όπως είπε και ο κύριος Ντεγκράντες ως Κιώδης, το θέμα του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, είναι κάτι το οποίο είχε συζητηθεί μετά από τις αρχικές αντιδράσεις των εμπλεκομένων φορέων. Θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στην περίπτωση τεχνητών λύσεων ή διευθετήσεων. Τώρα, αν υπάρχουν εναλλακτικές ε, λύσεις ή προτάσεις, θα μπορούσαμε και εμείς να συνδράμουμε για να δούμε ακριβώς τι προβλέπει ο νομοθέτης. Θα ήθελα επίσης να αντιδράσω στην πρόταση του σχεδίου σε σχέση με ε, την οικονομική δραστηριότητα στην χώρα παροχής των υπηρεσιών, δηλαδή στη χώρα προορισμού. Αυτό το θέμα μας απασχόλησε επίσης λεπτομερώς την Επιτροπή, έτσι ώστε η πρόταση να επιτρέψει σε επιχειρήσεις να μετακινηθούν στην εσωτερική αγορά, να εκμεταλλευτούν αυτή τη δυνατότητα δηλαδή, αλλά να μην υπάρχουν καταχρήσεις, να υπάρχουν δικλίδες ασφαλείας. Γι' αυτό Είπαμε και εμείς ότι καμία μετατροπή δεν θα πρέπει να επιτραπεί μέσα στα πλαίσια μιας ε, τεχνητής διευθέτησης. Η εισηγήτρια μιλά για την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα της παροχής υπηρεσιών, στη χώρα προορισμού. Έχουμε συνεργαστεί εκ του σύνεγγυς με τις νομικές υπηρεσίες της Επιτροπής και θεωρούμε ότι ότι ε, ενδεχομένω να υπάρξει ένα συνενετικό σχήμα σε σχέση με την απόφαση Portwood του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τώρα, σε σχέση με τη συμμετοχή των εργαζομένων, θα πρέπει να σας πούμε ποιο είναι το σκεπτικό μας. Δηλαδή να χτίσουμε πάνω στο κεκτημένο μέσα στα πλαίσια της οδηγίας, ε, της οδηγίας για τις ε, διασυνοριακές συγχωνεύσεις και ιδιαίτερα εκεί όπου κρίναμε ότι χρειάζονται περισσότερες διασφαλίσεις. Χαιρόμαστε γιατί η συγγήτρια έκανε πιο φιλόδοξες προτάσεις, αλλά να είμαστε και προσεκτικοί. Εμείς είμαστε πιο μετριοπαθείς στις προτάσεις μας σε σχέση με την συμμετοχή των εργαζομένων, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα στα κράτη-μέλη ως προς τη συμμετοχή των εργαζομένων. Και είναι δύσκολο να φτάσουμε σε έναν συμβιβασμό με τον άλλο νομοθέτη. Και ένα τελευταίο σημείο που κρίναμε άκρος ενδιαφέρον. Εσείς προτείνατε να έχουμε περισσότερες δικλίδες ασφαλείας σε σχέση με τον ε, διορισμό των ε, ε, διευθυντικών στελεχών και την ευθύνη που φέρουν. Αυτό το συζητήσαμε και στην προηγούμενη έκθεση σε σχέση με την αφαίρεση των δικαιωμάτων των ε, διευθυντικών στελεχών εκεί που επιβάλλεται. Θα πρέπει να ε, βρούμε συγκεκριμένες συνέργειες μεταξύ των δύο προτάσεων για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νίμπλα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια τον σκιώδη μας. Συμφωνώ και εγώ ότι η έκθεση αυτή εμπλουτίζει την πρόταση της Κομισιόν. Βεβαίως ακούστηκαν πολλές ιδέες, τις οποίες πρέπει να τις ε, εξετάσω. Πώς το είπατε, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, αξιολογητές, τρίτη. Θα πρέπει να το σκεφτώ τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει κάτι τέτοιο δεν είμαι και πολύ εξοικειωμένη λόγω του ότι γνωρίζω καλύτερα το γερμανικό δικαιικό σύστημα. Ένα ερώτημα ε, έχω να θέσω ωστόσο. Το είπα και στην έκθεση Ισγεύκα. Για μένα σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η απλοποίηση, η αξιοποίηση των ψηφιακών διαδικασιών κτλ. κτλ. Δεν θέλω όμως να περιοριστεί η αρχή ε, της ε, προφύλαξης. Και γι' αυτό Επαναλαμβάνω και εδώ ότι στο σύστημα της Γερμανίας οι συμβολεογράφοι έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, ρόλο που σε άλλες χώρες επιτελούν τα δικαστήρια, για παράδειγμα. Θέλω όμως ε, να εξασφαλίσουμε και αυτή τη διάσταση ε, όσον αφορά τις ψηφιακές διαδικασίες και να δούμε πώς μπορεί να ενταχθεί κάτι τέτοιο ε, στην, στην έκθεσή σας. Είπατε μετά για, για την... Ε, για την αποχώρηση κάποιου μετόχου. Εδώ υπάρχει άρθρο 86, παράγραφος 3, της Οδηγίας για την Κινητικότητα. Εκείνος που αποχωρεί, προβλέπεται εκεί, ότι θα πρέπει να το κοινοποιεί αυτό ηλεκτρονικά και μόνο. Εδώ θα ήθελα και η Κομισιόν και η εισηγήτριά μας να, να μας πούν πώς αξιολογούν αυτή τη διάταξη. Γιατί αυτό συνάδει με τους στόχους μας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε καλύτερα να διαγραφεί αυτή η πρόβλεψη ε, για λόγους ε, διαφάνειας, προκειμένου να είναι σαφές ε, ποιοι και τι μερίδιο έχουν σε μια εταιρεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Αυτά. Αν θέλει η κυρία Ρέγνερ, έχει το λόγο, ναι. Πολύ σύντομα. Βλέπετε κύριε Πρόεδρε ότι έχουμε εισέλθει στο ουσιαστικό μέρος της συζήτησης πλέον. Θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση βεβαίως και με τους Κιώδης και με την Κομισιόν. Πολύ σύντομα λοιπόν θέλω να πω τα εξής. Κύριε Ντεγκράντε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η νομική αβεβαιότητα που υπάρχει πρέπει να καταπολεμηθεί, πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Και σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας αυτό. Και να πω στην κυρία Νίμπλε ότι ακριβώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και που με ενδιαφέρει και εμένα. Πρέπει να, να δούμε τις λεπτομέρειες. Γιατί το πακέτο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ε, προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις, για τους εργαζόμενους, αλλά θα, για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει καλά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τις ε, λεπτομέρειες του θέματος. Όσον αφορά τους νομικές, νομικούς ε, εμπειρογνώμονες που αναφέρατε, εγώ δεν έχω κάποια οριστική τελική θέση αυτή τη στιγμή. Έχω την, τη θέση που εκφράζω και μέσα από τις τροπολογίες μου διδασκόμαστε και εμείς στην πορεία. Θέλουμε οι εμπειρογνώμονες μας αυτοί, ε, οι εμπειρογνώμονες αυτοί να είναι μάγοι, πρέπει να τα ξέρουν όλα. Θέλουμε να δούμε πώς αυτά θα εκφραστούν στην καθημερινή ζωή ε, μέσα στις επιχειρήσεις. Είμαστε ανοιχτοί όμως στη συζήτηση και όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα. Εγώ θέλω να τονίσω ότι εμείς είμαστε νομοθέτες. Και πρέπει να σας πω ότι οι αποφάσεις του δικαστηρίου πολλές φορές ε, κινούνται ακόμη και σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Στόχος μας, δικός μας, είναι να καταλήξουμε σε ένα συγκεκριμένο κανόνα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στις ηλεκτρονικές διαδικασίες να εξασφαλίζεται ότι τα πάντα θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως είναι στην πραγματική ζωή, έτσι να είναι και ηλεκτρονικά. Όσον αφορά αυτό που αναφέρατε κυρία Νίμπλερ για τους ε, μετόχους, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας ε, δώσω μια απάντηση. Θα το ελέγξω όμως το θέμα, θα το συζητήσω και θα, και θα επανέλθω. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και κλείνουμε το θέμα αυτό και συνεχίζουμε με το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Η είμαι εγώ. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το εξετάζουμε από κοινού με την Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων. Είναι ένα πολύ επίκαιρο και σημαντικό ζήτημα. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπη. Οι ε, συντονιστέ τη επιτροπή μα πριν από τι τερινές διακοπέ, αποφάσισαν να εκδώσουμε μια γνωμοδότηση προ την ΑΦΚΟ με την μορφή επιστολής και οριστικά εγώ συγητής το προσχέδιο θα διανεμηθεί. Ζητώ συγγνώμη πως μπορείτε να κάνετε λίγη ησυχία παρακαλώ. Θα προετοιμάσω λοιπόν ένα προσχέδιο κειμένου το οποίο θα διανεμηθεί μεταξύ των συντονιστών προκειμένου να συμφωνήσουμε επί αυτής της επιστολής. Η, ε, το προσχέδιο της έκθεσης της ΑΦΚΟ μας ε, κοινοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα και συνοψίζει τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν για το μέλλον της Ευρώπης ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να δώσει διευκρινήσεις και κατευθείαν γραμμέ για την κατεύθυνση την οποία μπορεί να πάρει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εν ώψη των εκλογών του 2019. Ο στόχος της έκθεσης δεν είναι λοιπόν να αποφασίσουμε επί διαφόρων λακτικών λύσεων, αλλά να ορίσουμε τα προβλήματα, να περιγράψουμε τις προκλήσεις και τις ενδεχόμενες ε, ε, λύσεις ή επιλογές που μπορούμε να έχουμε που θα έχουμε στην επόμενη θητεία. Η έκθεση της ΑΦΚΟ εστιάζεται στις βασικές προκλήσεις που, αντιμετωπίζουν, που αντιμετωπίζει το θεσμικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετανάστευση, την κρίση του ευρώ, το Brexit, ο προστατευτισμός και η εμπορική πόλεμη, η τρομοκρατία, η κυβερνοασφάλεια, η φοροαποφυγή, η προστασία των δεδομένων και άλλες. Εμείς ε, λοιπόν θα πρέπει να αναζητήσουμε προκλήσεις για το μέλλον της Ευρώπης στη δική μας αρμοδιότητα. Για παράδειγμα, αναλογικότητα και επικουρικότητα, η εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, καλύτερη νομοθέτηση και απλοποίηση, ε, δικαστική συνεργασία και τα νομικά και ηθικά ε, ε, ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Τα νομικά λοιπόν αυτά κυρίως θέματα θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στις προκλήσεις της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες και χωρίς να προτείνουμε ενδεχομένω λύσεις. Θέλουμε να τα περιγράψουμε, να περιγράψουμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες τα επόμενα χρόνια εν ώψη των εκλογών του 2019. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας πείτε τη, τη γνώμη σας. Και εγώ θα τη λάβω υπόψη μου κατά τη σύνταξη της επιστολής έκθεσης που θα ετοιμάσω. Ο κύριος Λεμπρετών θέλει το λόγο. Έχετε το λόγο κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι πολύ χρήσιμο ο προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης, το αναγνωρίζω. Αλλά είναι δύσκολο όταν το κείμενο παίρνει πολύ συγκεκριμένε ε, κομματικές θέσει θα έλεγα. Υπάρχουν κάποια καλά βέβαια. Η αναφορά στο Brexit, η αναφορά στο Λευκή Βίβλιο της Κομισιόν για το μέλλον της Ευρώπης, ασφαλώς. Αλλά τα υπόλοιπα... Ε, υπάρχει μια ικανοποίηση για τον εαυτό μας ότι έχουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παίξει το σημαντικό ρόλο για την ευημερία και την ειρήνη. Εντάξει, την ειρήνη ναι, αλλά η ειρήνη έχει πολλά αιτία και σίγουρα δεν είναι το μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι διαφορά την ευημερία, πρόκειται για μια δήλωση που θα πρέπει να τη δούμε, να τη σχετικοποιήσουμε. Εξαρτάται για ποιους μιλάμε, ποιους λαούς, ποια κομμάτια του κόσμου ε, δεν ευημερούν όλοι. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο απαξιώνει αυτό το κείμενο τη συζήτηση. Και μετά, λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ, διότι μετά τα τελευταία αποτελέσματα εκλογικά αποτελέσματα και μετά τις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές πριν από πέντε χρόνια εγώ θα φανταζόμουν ε, ότι θα είχε κάποιος ότι θα είχαν καταλάβει οι θύνοντες πως ε, ο κόσμος δεν θέλει ένα υπερκράτος ένα τέτοιου είδους μηχανισμό κι όμως η έκθεση τι κάνει προσθέτει και άλλα επίπεδα ε, ε ακούγεται, το διαβάζω σαν το χειρότερο ομιλία του πρόεδρου Μακρόν και ο κύριος Μακρό είναι εξαιρετικά φιλοευρωπαίος. Ε, κατανεμημένη κυριαρχία. Τι θα πει κυριαρχία κατανεμημένη, πώς είναι να τον αυτά είναι αντίφαση. Ε, δεν, ε, ή την έχουμε την κυριαρχία ή ε, την απαρνούμαστε αλλά δεν είναι δυνατόν να τη μοιραστούμε. Μπορούμε να μοιραστούμε αρμοδιότητες αλλά όχι κυριαρχία. Είναι παράλογο αυτό που λέει η έκθεση. Σημείο 5. Η υποκατάσταση, η αντικατάσταση μάλλον τις ε, ε με την ισχυρή πλειοψηφία, με την ισχυμένη πλειοψηφία. Το αντίθετο θα πρέπει να γίνει. Τρίτο παράδειγμα, σημείο 8, η μετατροπή του Συμβουλίου σε μια πραγματική νομοθετική, σε ένα πραγματικό νομοθετικό όργανο. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της προσδοκίας του λαού των λαών. Σημείο 14. Δημιουργία ενός Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Πρόκειται για μια πονδιοποίηση της Ευρώπης. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο δεν θέλουν οι λαοί. Είναι σαν να προκαλείτε τον Ταύρο με ένα κόκκινο πανί. Και μετά η γενίκευση των Spitzenkandidaten, των ε, ε, προέδρων, των, των επικεφαλής υποψηφίων και τέλο, το κερασάκι στην κούρτα ε, όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό, ενιαίο ευρωπαϊκό λαό. δεν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό λαό, υπάρχουν πολλοί ευρωπαϊκοί λαοί που είναι πολύ χαρούμενοι που διαφέρουν μεταξύ του και εγώ χαίρομαι που υπάρχουν τόσοι ευρωπαϊκοί λαοί δεν είναι δυνατόν αυτό αυτή η κατάσταση να αντικατασταθεί από ένα είδο εναρμονισμένου, μια είδους εθνική αρμονία που θα ε, βασιλεύει στην Ευρώπη. Ε, τι να σας πω. Καλό κουράγιο. Εγώ αν ήμουν εισηγητής θα προσπαθούσα να τα γράψω ξανά όλα από την αρχή. Δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Καλή, καλό κουράγιο. Well, thank you very much, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Λεμπρετών. Ευχαριστώ που μου εύσχεστε καλή επιτυχία. Με εκπλήσει η έκπληξή σας γιατί τα σημεία που θίξατε ε, φαίνονται σαν κάτι το καινούριο. Όμως το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και δύο χρόνια ενέκρινε τις εκθέσεις Μπρεσό Μπροκ ή την έκθεση Φερχόφστατ όπου αυτά τα σημεία είχαν γίνει αποδεκτά από την πλειοψηφή. Άρα δεν είναι κάτι το νεωτερικό. Σας ευχαριστώ όμως που μου εύχεστε τα καλύτερα. Τη στιγμή που δεν ε, ζητά κανείς άλλο το λόγο, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουμε με το θέμα υπαριθμών 12. Η εξέταση εξέταση της ευθυγράμμισης των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων στον τομέα της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής. Δυστυχώς η συγγήτρια, η κυρία Χάουταλα, δεν είναι μαζί μας σήμερα, άρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ανακοινώσω ότι η, υποβολή, η προθεσμία των τροπολογιών ε, έχει οριστεί στις 7, στις 7 Σεπτεμβρίου. Θέλετε το λόγο παρακαλώ. Εντάχει, παρά το γεγονός ότι η συγγήτρια δεν είναι παρούσα, θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε αυτόν τον κανονισμό ε, ώστε να υπάρχει σωστή κοινοποίηση των μέτρων για να υπάρχει καλύτερη διαφάνεια και υπάρχει υποχρεωτική λογοδεσία για τις 10 οδηγίες που έλαβε υπόψη η Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες προς το κοινό και προς την Επιτροπή και τα δεδομένα αυτά θα πρέπει να διατίθενται επιγραμμικά, να είναι δημόσια δηλαδή και να μην συντάσσονται στο χαρτί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Χάουταλα για ορισμένες από τις τροπολογίες της και χαίρομαι γιατί ζήτησε πιο ε, αποδοτική διαδικασία διαδικασία λογοδοσίας της Επιτροπής, ιδιαίτερα σε σχέση με την περιβαλλοντική πολιτική, μέχρι τον, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο και μετά κάθε τρία χρόνια. Να υπάρχει αυτή η διαδικασία λογοδοσίας. Όμως δεν κατανοώ γιατί η Επιτροπή στη νέα πρόταση δεν έχει υποβάλει νέες υποχρεώσεις σε σχέση με ζημίες στον τομέα του περιβάλλοντος και διαγράφεται το άρθρο 14.2. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή θα ήθελε να απαντήσει στην ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, γιατί μου δίνετε το λόγο και ακόμα και ρήμην της εισηγήτριας θα θέλαμε να την ε, ευχαριστήσουμε για την εργασία της αυτή την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε την ε, ε, βουλευτή που μίλησε υπέρ αυτής της νομοθετικής πρότασης και θα ήθελα να υπενθυμίσω γενικότερα ότι αυτή η νομοθετική πρόταση είναι από το ε, μίας ε, διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε πέρσι σε σχέση δηλαδή με την διαδικασία λογοδοσίας δυνάμει του περιβαλλοντικού δικαίου. Θέλουμε λοιπόν για 10 θέματα περιβαλλοντικού δικαίου να υπάρχει διαδικασία reporting και Τη στιγμή που υπάρχει άλλη διαφορετική νομοθεσία που δεν καλύπτεται από την τρέχουσα, τότε να το βλέπουμε κατά περίπτωση. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και τις παρόμοιες αλλαγές εκεί που υπάρχουν. Θέλουμε να προβάλλουμε ε, μία ε, μετατροπή υποδείγματος μία μετάβαση υποδείγματος σε σχέση με αυτά που ίσχυαν εδώ και 30 χρόνια, όπου οι πληροφορίες ε, ε, μεταφέροντας την Επιτροπή επί χάρτου με καθυστερήσεις ε, και φυσικά και η Επιτροπή καθυστερούσε στη συνέχεια. Και αυτό σε σχέση και με την δική μας λογοδοσία προς εσάς και το Συμβούλιο. Θα θέλαμε να ε, τονίσουμε ότι οι πληροφορία στον τομέα του περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για τους ε, πολίτες και αυτό αφορά και τις ε, τοπικές αρχές και κοινότητες. Επίσης, θα θέλαμε να κόψουμε τον διοικητικό φόρτο και τις επικαλύψεις, γι' αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να αυξήσουμε την διαφάνεια, να γίνει εξυγχρονισμός με τα νέα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και επίσης να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο. Θα ήθελα να μιλήσω για δύο πτυχές που προβλέπονται και από τις τροπολογίες. Καταρχήν θα θέλαμε οι βάσεις δεδομένων να ε, είναι επικαιροποιημένε για τη χρήση από το κοινό και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δηλαδή να μην ε, έχουμε ε, πεπαλαιωμένες πληροφορίες οι οποίες προβάλλονται στο κοινό και στα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό θα θέλαμε να έχουμε επικαιροποιημένες πληροφορίες από τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μην βασιζόμαστε σε ε, κοινοποίηση δεδομένων επί χάρτου. Και αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο αυτές οι αλλαγές θα ε, μειώσουν τη διαδικασία ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι ε, δεν πλήττονται οι ε, δικαιοδοσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την επικαιροποίηση αυτής της διαδικασίας, διότι τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα και Φυσικά η Επιτροπή θα λογοδοτεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό δεν θα θέλαμε να έχουμε μία περιοδική τριετή αναθεώρηση των διαφόρων ε, μερών της νομοθεσίας. Θεωρούμε ότι αυτό δεν συμβαδίζει με αυτά που θα μπορούσαν να γίνουν. Η αναθεώρηση αυτή χρειάζεται κατά μέσο όρο δύο χρόνια. Γι' αυτό αν γίνεται κάθε τρία χρόνια τότε αντικαθιστούμε ένα βάρος με ένα άλλο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ διότι διευκολύνεται αυτή τη διαδικασία και με χαρά να συνεργαστούμε με τον εισηγητή. Ευχαριστούμε και εμείς. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το θέμα και συνεχίζουμε με το σημείο 4. Εξέταση σχεδίου έκθεσης σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ο κύριος Τζαμπάσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Έπειτα από την πρόταση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο το Φεβρουάριο του 2018 η Επιτροπή μας επιφορτίστηκε με το καθήκον να συντάξει μια γνωμοδότηση. Ο κύριος Γιούγκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης συμπεριέλαβε για πρώτη φορά αυτήν την ιδέα της, της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας η οποία θα ενίσχυε τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και θα διευκόλυνε την ε, κινητικότητα των εργαζομένων. θα άνοιγε το δρόμο σε διασυνοριακούς κανόνες και θα υποστήριζε την ε, κοινωνική κινητικότητα στην Ευρώπη για εργαζομένους, για υπαλλήλους, για αυτοαπασχολούμενους, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για πολίτες τρίτων χωρών που νομίμως διαμένουν στην Ένωση. Η αρχή αυτή θα επιφορτιστεί κατά κύριο λόγο με την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και την οικοδόμηση ε, εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με απότερο στόχο όχι απλώς την κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά τη δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων. Μέσω αυτής της ενιαίας θηρίδας, λοιπόν, θα συγκεραστούν οι διοικητικές ε, ικανότητες και δυνατότητες ε, πολλών ευρωπαϊκών αρχών. Όσον αφορά την έκδοση ε, καρτών εργασίας, καθεστώτων ασφάλισης, την επίλυση διαφορών, διαφορών μεταξύ εθνικών αρχών ή διαφορών που σχετίζονται με καταγγελίες παραβίασης της νομοθεσίας, ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας ή την αδήλωτη εργασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ άλλων τονίζει ότι σε καμία περίπτωση η διαδικασία αυτή δεν θα επιβαρύνει διοικητικά τα κράτη-μέλη, τους εργοδότες ή τους εργαζομένους. Ούτε θα επιφέρει κάποιες αλλαγές στην εθνική νομοθεσία τονίζει η Κομισιόν. Και είναι αποφασιστικής σημασίας το στοιχείο ότι θα εναπόκειται στη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών το αν και πώς θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που θα τους προσφέρει αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα σχετικά εχέγγυα που κατοχυρώνονται και στο δεύτερο πυλώνα μας οδηγούν ως κοινοβούλιο να τονίσουμε την ανάγκη προστασίας των εθνικών αρχών και στο κείμενό μου αναφέρομαι και σε κάποιες ανησυχίες που έχω εγώ και που θέλω να συζητήσω και μαζί σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τις ε, σημαντικές κυβερνοαπειλές που αντιμετωπίζουμε στον σύγχρονο κόσμο, το ρόλο των κρατών μελών, των κοινωνικών εταίρων, ιδίως όσον αφορά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτής της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Και τέλος, αναφέρομαι και στον, στη χρηματοδότηση αυτής της αρχής. Η Κομισιόν προτείνει σημαντικότατο προπολογισμό. Αλλά το από πού θα προέλθουν αυτά τα χρήματα είναι ακόμη άγνωστο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Ζάμιτ. Νομίζω πως ε, συζητούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πρόκειται για τις θεμελιώδεις ελευθερίας και μία από αυτές είναι η ελευθερία κίνησης. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να εργάζονται, να διαμένουν και να σπουδάζουν οπουδήποτε θέλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κινητικότητα του εργατικού δυναμικού όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνεται με πιο συντονισμένο και εναρμονισμένο τρόπο. Γι' αυτό το λόγο και είναι σημαντική η είδηση της Ευρωπαϊκής ε, Αρχής ε, ε, Εργασίας. Ε, υπάρχουν πολλά διασυνοριακά στοιχεία, κοινωνικά, θέματα κοινωνικών εισφορών, αποτελεσματικής εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ομαθησίας. Πολλά από αυτά είναι προβληματικά. Μάλιστα οι εργαζόμενοι μπορεί να ε, ε, ε, καταλήξουν σε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις, να μην μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους κλπ. Ενώ οι επιχειρήσεις μεταξύ τους μπορεί να υφίστανται αθέμητο ανταγωνισμό όταν δεν εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες παντού. Γενικότερα, τα θέματα μετανάστευσης χαρακτηρίζονται από έλλειψη υπαρκού προγραμματισμού. Για παράδειγμα, πολλές ε, φορές η αύξηση του εργατικού δυναμικού μιας χώρας είναι πολύ μεγαλύτερη από τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι φεύγουν για να δουλέψουν σε άλλη χώρα. Οπότε, Συμφωνώ και με πολλές από τις τροπολογίες που προτείνουμε και να σας υπογραμμίσω ορισμένε από αυτές. Ιδιαίτερω τροπολογίες οι οποίες αφορούν την προστασία των δεδομένων, μία, μάλλον περισσότερες τροπολογίες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμπλέκεται στη διαδικασία, διότι ο οργανισμός αναφέρεται στην Κομισιόν, αναφέρεται στα κράτη-μέλη, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αγνοηθεί. Θέλουμε όμως να είμαστε τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επίσης υπάρχουν τροπολογίες σχετικές με την πρόθεση των ευκαιριών εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άτομα ανάπηρα και ειδικές ανάγκες. Συνεργασία των κρατών μελών για θέματα επίσης ανταλλαγή, διασυνορικής ανταλλαγής δεδομένων και εφαρμογή του νόμου. Επίση, αν η διαδικασία διαμεσολάβηση δεν δώσει αποτέλεσμα, πρέπει να είναι σαφέ ποιε νομικές, ποιες δικαστικές αρχές είναι υπεύθυνε. Τέλος, κανόνες ε, λογοδοσίας, διότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτή η αρχή, αν ιδρυθεί, θα λογοδοτεί σωστά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Ευχαριστώ πολύ όλα τα, για όλα τα σχόλια. Μέσω αυτής της αρχής μπορεί πράγματι να βελτιωθεί πολύ κατά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν είχε πρωτοανακοινωθεί αυτή η ίδρυση, είχα σκεφτεί πως αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε κίνητρα στους νέους να σπουδάζουν στο εξωτερικό, να ε, κάνουν εθελοντισμό, ε, να μετακινούνται περισσότερο και θα πρέπει να στηρίξουμε ε, όλους όσοι είναι φορείς που στηρίζουν την κινητικότητα. Έχουμε δει στο παρελθόν εργαζόμενους οι οποίοι κινούνται διασυνοριακά, αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα και στην κοινωνική ασφάλιση και στην ασφάλιση υγείας, αργότερα στη σύνταξή τους, όταν συνταξιοδοτηθούν, ακόμα και σε ζητήματα τραπεζικών λογαριασμών υπάρχουν προβλήματα διασυνοριακά. Εμείς με αυτή την αρχή μπορούμε να συνεισφέρουμε στο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Ακόμα και στις ε, Ακόμα και εκεί που υπάρχουν κανόνες, όπως για παράδειγμα στις ε, συνοριακέ περιοχές, μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν στους συναδέλφους που έχουν αναλάβει το θέμα αυτό Ας περιμένουμε την ψηφοφορία έτσι ώστε η Ευρώπη να δώσει ένα θετικό μήνυμα πριν τις επόμενες εκλογές. Κύριε Ρέγνερ, είναι σημαντικό η αρχή να είναι αρχή, πραγματική ευρωπαϊκή αρχή, να μην περιοριστούμε στη διαμεσολάβηση. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ πρακτικοί και ρεαλιστές. Έχουμε εμπειρία σε, ευρωπαϊκό, εθνικό επίπεδο. Όταν εντοπιστούν παρατυπίες σε ένα έλεγχο μιας επιχείρησης, για παράδειγμα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, μια αρχή, μια αρμόδια αρχή απευθύνεται στην ομόλογή της σε, άλλο, σε άλλη χώρα, εκεί από όπου προέρχεται για παράδειγμα ο προκειμένου να του χορηγηθούν τα δικαιώματά του, αλλά αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει όλα μπορεί να θαυτούν σε κάποιο σιρτάρι. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά υπάρχουν εθνικοί μηχανισμοί πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους πολλές φορές και αυτό οδηγεί στη λύθη, οδηγεί στην δημιουργία εκκρεμών υποθέσεων που δεν λύνονται ποτέ, που δεν δίδεται συνέχεια ποτέ σε αυτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν κανόνες που θα οδηγούν σε ελέγχους και που θα εφαρμόζονται. Χρειάζεται λοιπόν μια ευρωπαϊκή υπηρεσία όπως κάναμε και με τις τράπεζες. Και ήδη είχαμε καθυστερήσει με τις τράπεζες. Όμω είδατε πω η νομοθεσία βοήθησε στον τραπεζικό τομέα. Ευχαριστώ, κ. Λεμπρετό. Oui, merci, Monsieur le Président. Je, suis désolé de briser une fois de plus le consensus qui est. <laughs> Ζητώ συγγνώμη που διακόπτω αυτή την συνένεση. Ε, οι, οι τροπολογίες και το κείμενο του ΣΥΓΙΤΗ ε, προσπαθούν να βελτιώσουν πράγματι το αρχικό κείμενο με τραβούν, με έλκουν ιδιαίτερα οι τροπολογίες ε, που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα ουσίας. Αυτή η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας είναι πραγματικά απαραίτητη. Θα μου πείτε ε, είσαι μειοψηφία. Όμως εδώ τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Πολλά εθνικά κοινοβούλια πιστεύουν αυτό πιστεύω και εγώ. Το τσεχικό, το πολωνικό και το σουηδικό κοινοβούλιο θεωρούν ότι παραβιάζεται η αρχή της επικορικότητας, ότι ε, ε, υπησερχόμαστε σε εθνικές πολιτικές, όπως η πολιτική για την κοινωνική ασφάλεια, ασφάλιση. Τροπολογίες οι οποίες προτείνει ο εισηγητής δεν μας αρκούν, δεν αρκούν στην ομάδα μου για να ψηφίσουμε υπέρ δεν μπορούμε να δεχτούμε την ίδρυση αυτής της αρχής, η οποία κατά την άποψή μας είναι περιττή, γραφειοκρατική, δαπανηρή. Και πιστεύουμε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να απαντήσει στις προσδοκίες των λαών της, να εστιάσει στα σημαντικά και όχι να προσπαθεί να ροκανίσει εθνικές αρμοδιότητες. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε λοιπόν και αυτό το σημείο, εκτός και αν θα ήθελε κάτι να προσθέσει ο εισηγητής, φαίνεται πως όχι, άρα τελειώνουμε και με το σημείο υπαριθμών 4. And we will now proceed by... Και στη συνέχεια θα ψηφίσουμε Παρακαλώ να έχετε έτοιμες τις κάρτες σας. Before we start voting, πριν αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι για τα σημεία 17 και 18 θα συνεχίσουμε τις ψηφοφορίες ε, και κλεισμένων των θυρών και γι' αυτό θα γίνει ένα διάλειμμα για να είμαστε σε σύνθεση και κλεισμένων των θυρών.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 δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε υπεράριθμους από το ΕΛΚ ένα ή δύο. ΟΚ ΟΚ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 It seems that we can... Ωραία, φαίνεται ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν για την τυθάσευση της παγκοσμιοποίησης, ε, εμπορικές πτυχές, σχέδιο γνωμοδότησης ε, του κυρίου Λεμπρετών. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ να γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Εγκρίνεται. 10 προς 9. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά sorry, sorry. Oh, sorry. Uh, clearly adopt. Σαφώς εγκρίθηκε. Τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, παληθεύουμε ηλεκτρονικά. και εγκρίνεται. 16 υπέρ. 16 υπέρ κατά. Αποχές. Με συγχωρείτε πρέπει να επαληθεύσουμε για άλλη μια φορά. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 34 απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά. Ελέγχουμε την 36 παρακαλώ. Εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Και τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί του σχεδίου γνωμοδότησης. Εγκρίνεται. Να συγχαρούμε λοιπόν τον κύριο Λεμπρετόν. Συνεχίζουμε με την αναδιοτύπωση σε σχέση με την χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα. Η κυρία Γκέριγκερ είναι η συγγήτρια. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά αρχιτεί ψηφοφορία. Ε, εγκρίθηκε. Να συγχαρούμε την κυρία Γκέριγκερ. Και συνεχίζουμε με την αναδιατύπωση σε σχέση με τους οργανικούς ε, ρήπους. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, έκθεση Γκέριγκερ. adopted and now comes the και τώρα διακόπτουμε γιατί η νέα ψηφοφορία θα γίνει, η επόμενη μάλλον θα γίνει και κλεισμένων των θυρών. Γι' αυτό όσοι δεν πρέπει να παρίστανται να αποχωρήσουν παρακαλώ.